Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λέει η Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αρχίζουμε να έγκριση της ημέρησης διάταξης και σας ενημερώνω ότι ζητήθηκε αλλαγή για την ημερήσια διάταξη. Ανάλογα με το ποιος μπορεί και δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Οπότε τα σημεία 4 και 5 θα αντιστραφούν, η σειρά που θα τα εξετάσουν δηλαδή, θα αντιστραφεί δηλαδή το θέμα της ε, Παγκοσμίου Τράπεζας θα ζητηθεί πρώτο και κατόπιν θα συζητήσουμε την πρόταση για το CPR. Συμφωνείτε? Ωραία. Και με αυτή την αλλαγή εγκρίνεται την σε διάταξη. Ανακοινώσει τη Πρόεδρου δεν έχουμε και τόσο πολλέ. Απλώ το ότι είχαμε μια πολύ πετυχημένη αποστολή στην Σλοβενία. Πάθα θα μας τα πει όμως καταλεπτός ο κύριος Φανιθελόη αργότερα. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 3 της ενεργητικής διατάξεως και πρόκειται για την ε, συζήτηση του σχεδίου νομοδότησης για την αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στήριξης διαρροτικών μεταρρυθμίσεων πρώτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά για την προσαρμογή του γενικού του στόχου. Η κυρία Ρούζα Τόμασιτς είναι η συγγετρία. Έχει γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και έχουμε το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες και τις ψηφοφορίες όσον αφορά το κείμενο. Οπότε να δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Τόμας και θα συνεχίσουμε με τους σκιώδες συζητητές και τα μέλη της Επιτροπής μας. Κυρία Τόμας, ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας τα πω στα κροατικά. Στις 20 Μαΐου 2017 το πρόγραμμα στις διεργασίες μεταρρυθμίσεων τέθηκε σε ισχύ για την περίοδο 17 έως και 20. 142,8 εκατομμύρια ευρώ είναι περικοδότηση και αυτό θεσπίστηκε ούτω ώστε να υποστηριχτούν οι δυνατότητε των κρατών μελών για να προτιμάσουν και να υλοποιήσουν και τι δικέ μεταρρυθμίσει ε, προς όφελος της ε, ανάπτυξης και μέσω κάποιας ε, αρρωγής, τόσο ώστε να υπάρχει αποτελεσματική απορρόφηση των κοινωνικών κονδυλίων. Εμείς συμφωνήσαμε στην προσπάθεια να βοηθούν τα κράτη-μέλη για διάφορες πολιτικές. Έχει καταδείξει η εμπειρία ότι πολλά κράτη-μέλη ζητούν βοήθεια για το πρόγραμμα και αυτό αφορά όλες τις ε, πολιτικές που καλύπτονται Φερρυπίν, διακυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, διαχείριση των εσόδων, των δημοσιονομικών, επιχειρήσεις, απασχόληση, παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια, χρηματοοικονομικά και πρώτα στη χρηματοδότηση είναι σημαντικό το ότι το πρόγραμμα αυτό δεν επικαλύπτονται με άλλα προγράμματα. Μόνο όπου δίνει προσθεμένη αξία λειτουργεί. Και μαζί με εμπειρογνώμονες θα διατεθεί στα κρατη για τα έργα και σχέδια προετοιμασίας. Όλα αυτά θεωρούμε ότι έρχονται στη σωστή στιγμή και δημιουργούν ε, προσθέμενη αξία και ότι βοηθούν τα κρατη Οπότε και γι' αυτό δεν μας ε, εκπλήσει το τα κράτη-μέλη δείξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τόνιζα στην έκθεσή μου ότι είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των αρχών εταιρική σχέσης και θα πρέπει να εμπλακούν κοινωνικοί εταίροι και κοινότητα των πολιτών. Όταν έρθει η ώρα να αποφασιστεί ποια θα είναι η ακολουθητή στρατηγική επίσης και για τη διαδικασία εποπτείας κατά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, τη σωστή εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, έλαβα υπόψη μου το ότι η αύξηση της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος θα πρέπει να γίνει χωρίς να θυγούν άλλα σημαντικά ταμεία ή κονδύλια για τα κράτη-μέλη έχουν δικές τους πρωτοβουλίες. Το SRSP, θεωρείται ότι είναι το πιο δόκιμο μέσο σε σχέση με τις συστάσεις για την κάθε χώρα. Διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή, στις υπηρεσίες, στην ποιότητα διοικητικών και δεσμευμένων υπηρεσιών, σε δημόσιες υπηρεσίες και για την βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να προσαρμοστούν στα όσα ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, να υπάρξει επίσης δημοκρατική νοημοποίηση και να μην υπάρξει η ίδια προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη. Επομένω, το, το μέσο βελιξή είναι ο μόνο τρόπο τόσο να υπάρξει κάποιο είδου τέτοια, τέτοια του προγράμματο. Και έχουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάση των διορθωτικών ε, και τεπεντικών ταμείων γιατί είπαμε στην περίοδο μέχρι το 2020 δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει κάποιο μεταφορά κονδυλίων στο πολιτές δημοσίου πλαίσιο μόνο με αναθεώρηση αυτού και θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιηθεί το απόθεμα ε, κατεπήγοντος και θα πρέπει να δούμε τι μέσα προβλέπει ο κανονισμός του MFF, οπότε είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το μέσο ευελιξίας είναι η μόνη επιλογή για την ε, χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για το πρόγραμμα, για ό,τι δυνατότητες, για όλες τις που ε, προσφέρονται, τόσο ώστε όλοι να μπορούν να προετοιμαστούν για τα σχέδια και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το εθνικό συμφέρον και τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε θέλουμε να κάνει ενημέρωση η Επιτροπή στα κράτη-μέλη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Κροατικά. Οπότε και εγώ περιμένω την συνεργασία μαζί σας, τις προτάσεις σας, για να μπορέσουμε με επιτυχία να ολοκληρώσουμε αυτή την γνωμοδότηση και τα κατημέλη να, τη, να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, να υποβάλουν τις προτάσεις τους τον Οκτώβριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέσο πολιτικής. Πρέπει να αποσπάσουν λοιπόν αποτελέσματα με την χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Να κάνουν τη σωστή χρήση αυτών και έτσι να γεφυρωθούν οι οικονομικές ανισότητες. Και τώρα έχουμε τη, την κυρία Μάλετης με τους κοιόδες ηγητές. Η κυρία Μάλετης. Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι πως οι δραστηριωτικέ μεταρρυθμίσεις χρειάζονται και πρέπει να εφαρμοστούν για να πετύχουμε καλύτερα αποτέλεσματα στην πράξη. Οι τροπολογίε μας όμως θα πρέπει να, δίνουν το εξής μήνυμα. Πρώτον ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για να ε, υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και για αυτή την πολιτική βούληση χρειάζεται συμφωνία και στήριξη διαφόρων τμήματων της κοινωνίας. Πρέπει δηλαδή οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να εμπλέκονται εξ αρχής το ίδιο και οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιστήμονες, και άλλες ομάδες του πληθυσμού. Αυτό και για να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα, τη σταθερότητα των, των μεταρρυθμίσεων. Γιατί αλλιώς θα χρηματοδοτούνται τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή η κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα είτε να εμπλέξει είτε να μην εμπλέξει ε, ομάδες πολιτών της κοινωνίας κλπ. Ας είμαστε πολύ σαφείς ότι είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα των μετακινήσεων πολιτική συμφωνία, πολιτική βούληση και συμφωνία από όλα τα μέρη της κοινωνίας. Λοιπόν, δεύτερον, Και αυτή η παρατήρηση μου έχει σχέση με τα αποτελέσματα που περιμένουμε να έχουν οι διασωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο στόχος μας είναι ο βέλτιστος συντονισμός των ειδικών πρακτικών, είναι να συνδέσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές με το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις αναχώρασης τάσης. Είναι στόχος μας να συνδέσουμε το κείμενο αυτό με τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να βελτιωθεί η απροφητικότητα. Η εισηγήτρια λέει ότι θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την πολιτική συνοχής αλλά η πρόταση ίσω δεν, δεν έχει ακριβώ την ίδια κατεύθυνση. Οπότε συμφωνούμε σε όλα, αλλά αυτό το εργαλείο είναι μικρό. Δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε, να θέσουμε προτεραιότητες. Και θέλω να σχολιάσω και το θέμα των κοινών διατάξεων με το απόθεμα αποδοτικότητας, ε, επίδοσης μάλλον. Ε, αυτές είναι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις σχετικές με την πολιτική συνοχής, οπότε ας εστιάσουμε στον οικονομικό συντονισμό, την οικονομική πολιτική, την ΟΝΕ και ας είμαστε σαφείς στο μήνυμά μας. Επίσης, άμα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της μεταρρυθμιστικής ατζέντα. Ας είμαστε ξεκάθαροι διότι αποφασίζουμε για το μέλλον. παρόλο ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το απόθεμα επίδοσης. Μετά, χρηματοδοτικές πηγές. Η Κομισιόν λέει θα χρησιμοποιήσουμε το όργανο ευελιξίας, το όχημα ευελιξίας που έχουμε, τα 80 εκατομμύρια, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ναι στο εργαλείο ευελιξίας και όχι στην τεχνική συνδρομή για την πολιτική συνοχής. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την πολιτική συνοχής σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με πολλούς άλλους τομείς. Οπότε ναι, στο διευκόλυνση ευελιξίας αλλά τελικά ποιο θα είναι το μήνυμα μας για το μέλλον. Πώς θα συνδεθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις με την πολιτική συνοχή, πώς θα χρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί έχουμε δει την πρόταση της Κομισιόν Έχουμε υιοθετήσει πολλές ε, εκθέσεις και εδώ και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Αλλά πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική συνοχή με αυτό το όργανο, με αυτό το εργαλείο. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, ε, αλλά από τώρα ας είμαστε σαφείς. Thank you very much. The next shadow rapporteur, Mrs. Krell. Η άλλη κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση πρώτα πρώτα, μια διασάφηση. Για ποιο πράγμα μιλούμε ακριβώς. Η πρόταση για τον μηχανισμό αυτό, SRSP, δηλαδή Structural Reform Support Program, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τις χώρες να επιφέρουν ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, το νόημα είναι, δεν θα κάνω εγώ, δηλαδή η Επιτροπή, τις μεταρρυθμίσεις αυτές για λογαριασμό σας, αλλά θα σας διαθέσω έμπειρο γνώμονες για να σας βοηθήσουν να κάνετε εσείς τις μεταρρυθμίσεις. Επομένως, μπαίνει στην τεχνική στήριξη στη τεχνική βοήθεια και γι' αυτό επιμείναμε εμεί όταν δίνουμε εμεί χρήματα, τα χρήματα αυτά πρέπει να έχουν σχέση με την πολιτική συνοχή. Τώρα, η πρόταση είναι διαφορετική, η οποία είναι πάντοτε μέλη δική μα αρμοδιότητα, αλλά η χρηματοδότηση πλέον δεν θα προέλθει από την τεχνική βοήθεια και η ΣΥΑ, και την ευχαριστώ, είπε ότι θα προέλθει από το μηχανισμό ευκαμψία, από το εργαλείο αν θέλετε ευκαμψία. Αυτό όμω με αυτόν τον τρόπο διαφεύγει πλέον, ξεφεύγει από την πολιτική συνοχή. Δεν δίνουμε πλέον εμεί χρήματα για την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό τονίζω να απομακρυνθούμε λίγο από την άμεση και άκαμπτη διασύνδεση με την πολιτική συνοχή, να είμαστε πιο εύκαμπτοι ώστε οι, Ευρωπα... οι χώρες μέλη με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν τη βοήθεια εμπειρογνώμων της Κομισιόν για τις διαδοτικές τους μεταρρυθμίσεις και η συνολική διαδικασία τελικώς να μην περιπλακεί έτη περαιτέρω. Διότι το νόημα δεν είναι να γίνουν τώρα δα οι μεταρρυθμίσεις, αλλά να δοθεί βοήθεια ώστε να μπορέσουν να κοιτάξουν ποιες είναι δυνατόν να γίνουν, ποιες όχι, ποιες είναι αναγκαίο να γίνουν, ποιες όχι. Γι' αυτό συνιστώ η διασύνδεση με τοπικές και περιφερειακές αρχές να μην διατυπωθεί τόσο αυστηρά. Εάν οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες ήδη με υποστήριξη εμπειρογνωμόνων, ε, για την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων μάλλον, να ρωτούν και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και αν θε, πρέπει να ρωτούν τις τοπικές περιφερειακές αρχές δεν χρειάζεται πλέον τους εμπειρογνώμονες. Τότε λοιπόν ολόκληρο το οικοδόμημα γίνεται άκαμπτο. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια για την πρώτη έκθεση του προγράμματος υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και όταν κάθισα να μελετήσω το πρόγραμμα, τότε άρχισα να καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Ο Λαμπέρ Βανίστερ Ρόι και εγώ, που είχαμε συνεργαστεί τότε, πήραμε κάποια απόσταση και είπαμε ναι, οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τις χώρες μέλη. Αυτές να αναλάβουν την διοργάνωση. Και βεβαίως κάθε χώρα μέλος έχει διαφορετικό σύστημα συμμετοχής κοινοβουλίων, ε, κοινωνικών εταίρων κ.ο.κ. Αλλά πρέπει να γίνει βέβαια καθαρή εργασία. Αυτό ναι. Δεν είναι όμως δικό μας ενδιαφέρον να προσθέσουμε και άλλα εμπόδια ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εν τέλει το SRSP. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό. Μία ακόμα παρατήρηση. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το παραφορτώσουμε βάζοντας μέσα και τις μελλοντικέ χώρες που ενδέχεται να ενταχθούν στη ζώνη ευρώ. Εδώ υποθέτω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στη διάρκεια του Μαΐου μαζί με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και στις 2 Μαΐου, 2, Μαΐου, ε, στις 2 Μαΐου ήδη ε, θα πει τα σχετικά. Δεν χρειάζεται να το εγγράψουμε στον δικό μας μηχανισμό. Θεωρώ ότι ο μηχανισμός που συζητούμε είναι αποτελεσματικός διότι βλέπετε καταναλώθηκαν τα κονδύλια. Θα ήθελα λοιπόν ο κανονισμός να είναι λιτός, απλός, με όσο δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα. Αλλιώς ενδεχομένως να, να, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι τον Οκτώβριο. Από ό,τι έχω καταλάβει, για την ώρα δεν υπάρχουν κονδύλια και όσο περισσότερο καθυστερεί το Κοινοβούλιο και μετά θα χρειαστούν και τριμερείς διάλογοι κλπ. τόσο περιπλέκεται η κατάσταση. Αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, καλύτερα να δείξουμε κάποια αυτοσυγκράτηση με κάποιες λίγες τροπολογίες τις οποίες προτείνει η συγκεντρία να συμφωνήσουμε με τον μηχανισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Τις συζητήσεις για την performance reserve θα την κάνουμε αμέσως τώρα σε λίγο. Και εκεί έχω ξεκάθαρη θέση, το γνωρίζετε. Μπορούμε όμως να τα πούμε μετά, θα είστε κι εσείς εδώ παρούσες και παρόντες. Εγώ νομίζω αυτόν εδώ το μηχανισμό να τον κάνουμε όσο, ξαναλέω, όσο πιο λιτό και ελαφρό γίνεται, χωρίς να επιβαρύνεται από πολλή γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ. Τώρα, Άλντε, ο κ. Γιακόφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κυρίες ε, Μάλετιτς ε, και Κέλ τα έχουν πει. Εγώ τώρα δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν, γι' αυτό και δεν θα μπω τόσο πολύ στο θέμα και στα επιχειρήματα που ακούστηκαν, με τα οποία άλλωστε συμφωνώ, αλλά θα μιλήσω για το τελευταίο αυτό που έδειξε η κυρία Κρέλ, δηλαδή την ε, εισαγωγή του ευρώ ως νομίσματος και την πολιτική γύρω από το ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να κάνουν οι χώρες εκτός ζώνης ευρώ για την ενίσχυση της οικονομίας τους κλπ, ανταγωνιστική οικονομία κλπ, μερικές στατιστικές μάλιστα δείχνουν καθαρά εκτός από Τσεχία, Σλοβακία και Σλοβενία, όλες οι άλλες χώρες μέλη, εννέα χώρες μέλη είναι αυτές, δεν έχουν ανταγωνιστικές οικονομίες. Σαφέστατα. Θα χρειαστεί λοιπόν να τους διατεθούν πολλά κονδύλια για ενίσχυση. Εγώ είμαι μεταξύ των οπαδών του κοινού νομίσματος ευρώ και θα ήθελα να μπορέσουν όλες οι χώρες μέλη να το υιοθετήσουν. Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν όμως σοβαρά μεταρρυθμιστικά μέτρα και βεβαίως και η σχετική χρηματοδότηση. Εγώ είμαι Κροάτης και γνωρίζω ότι η Κροατία θέλει το ευρώ. Άλλες χώρες μέλη δεν το θέλουν. Υπάρχουν όμως και άλλες που το θέλουν. Εάν τώρα ο Γιόνκερ δεν βγει να εξαγγείλει νέα στρατηγική για το ευρώ, κάτι το οποίο είναι και αυτό πιθανό, δεν θα είναι λάθος τότε στην περίπτωση αυτή νομίζω να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυτό, διότι εν τέλει ένα μέρος της πολιτικής συνοχής θα επηρεαστεί. Θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομία των χωρών αυτών, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα όσων θέλουν να επιτύχουν την εισαγωγή του ευρώ. Ξαναλέω ότι το ευρώ, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό και εκφράζω την ευχή και άλλες χώρες να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, συνάδελφό μου κυρία Ράιντκε που είναι η συζητήτρια για τούτο τον φάκελο. Μου έχει δώσει κάποια σχόλια να σας τα διαβάσω. Εμείς οι πράσινοι ενδιαφερόμαστε να εμποδίσουμε να πάρουν κονδύλια της πολιτικής συνοχής και να κλείσουν άλλες χρηματοδοτικές τρύπες και ειδικά για το SRSP, για το οποίο εμείς είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί, το έχουμε ξαναπεί. Η καλύτερη συμβολή σε οποιαδήποτε συνοχή είναι μια ξεκάθαρη και στέρεα πολιτική συνοχή με κονδύλια τα οποία θα τα κρατάει ίδια, δεν θα, επιτρέπεται να δίνονται σε άλλε πολιτικέ. Στο σχέδιο εκθέσεω υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία. Αφενό δηλαδή βασικανοποιούν οι προτάσει τη συγκίτρια για την ενίσχυση της αρχής ε, της ε, εταιρική σχέση και την συμμετοχή τοπικών περιφερειακών αρχών εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών κλπ. Όλα αυτά εμά τους πράσινους μας ενδιαφέρουν πολύ, τα βρίσκουμε πολύ σημαντικά και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν. Χαιρετίζουμε και την πρόταση για τον περιορισμό πρόσθετων κονδυλίων από τον μηχανισμό ευκαμψίας και κονδυλίων από την τεχνική βοήθεια. Αλλά αυτά τα απορρίπτουμε για το SRSP. Για μας τίθεται πολλές ερωτήσεις. Πώς θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια προγράμματα ή μάλλον ποια έργα θα υποστηρίξει και με ποιο τρόπο. Και ποια ιεραρχία, ποια προτεραιότητα θα δώσει σε προγράμματα. Θα βάλει ως κριτήριο τη συμμετοχή περιφερειακών αρχών. Δεν θα πρέπει όμως να είναι κριτήριο η ικανότητα συγχρηματοδότησης για να μπορέσουν να αποβληθούν τα κονδύλια αυτά. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, δεν βλέπω άλλον σκιώδη να είναι εδώ. Οπότε, για να δούμε μήπως κάποιος άλλος συνάδελφος άλλος Επιτροπής θέλει το λόγο. Όχι. Προς το παρόν, οπότε, έχουμε την ικανοποίηση να Καλώς ορίσουμε τους φιλοξενουμένους από την Επιτροπή των Περιφερειών και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τους ε, εισηγητές για το ίδιο θέμα στα θεσμικά του όργανα. Οπότε πρώτα-πρώτα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Όγκα Σίχεν, την ε, εισηγήτρια της Επιτροπής των Περιφερειών. Έχετε το λόγο κυρία. Merci, Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιφερειών στην συνεδρίαση και είχα την τιμή να ήμουν εισηγήτρια τη Επιτροπή των Περιφερειών τότε που ε, είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά η σχετική πρόταση αυτού του προγράμματος το 2016 και πότε το τότε γνωμοδοτήσαμε και εγκρίναμε στις 22 Μαρτίου το σχετικό κείμενο. Οπότε στηριζόμαστε σε αυτά τα αποθέματα, τόσο ώστε να έχουμε τις απαραίτητες διαρροτικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημόσιας δίκης σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Οπότε αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η μητέρα όλων των ε, μεταρρυθμίσεων, είναι προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 76% είναι αυτές οι συστάσεις, δηλαδή 59% για το 78% και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ και μια εδαφική διάσταση, ε, δηλαδή στηριζόμαστε σε τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές για την υλοποίηση. Οπότε ως επιτοπλίστων το θέμα είναι η ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων και έχουμε διατυπώσει κάποιες συστάσεις για αυτές τις δυνατότητες ε, για τα 25 κράτη-μέλη αλλά στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, ή περιφέρειες υπάρχουν προβλήματα. Οπότε και εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι πολύ θετικό και αυτό, αυτό το ΠΑΣ. Και είπαμε ότι υπάρχουν και κάποιες ε, προϋποθέσεις, οπότε ενισχύθηκε η θέση μας, οπότε προχωρήσαμε σε εταιρική σχέση με τα διάφορα επίπεδα ε, διακυβέρνησης της χώρας Ε, για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, μισό λεπτό υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Να βρούμε το κείμενο. Επίσης, ζητήσαμε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ ως εταιρική σχέση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης κάθε χώρα. Οπότε με ικανοποίηση είπαμε ότι αυτά όλα τα σωμάτων και στο δικό σας κείμενο. Επίσης ζητήσαμε την Επίτροπη το να θεσπιστούν κάποιε κατευθυντήρε, ούτω ώστε να υπάρχει συντονισμό για όλα τα μέτρα και τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό το ΠΑΣ θα έχει και συντονιστικό ρόλο. Όμω είπαμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί να μην έχουμε επικάλυψη και να μην έχουμε χρηματοδότηση τη ίδια δράση δύο φορέ. Επίση, ζητήσαμε το ΠΑΣ να δούμε τι θα γίνει με το 2020, να γίνει πρώτα μία αξιολόγηση για την επίδοση και όταν αυτό επιβιωθεί τότε θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσον υπάρχει συνοχή, ε, να δούμε πώς έχει λειτουργήσει και να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή των Περιφερειών. Άρα πρέπει να διαπιστωθεί ότι σήμερα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα γιατί η Επιτροπή δεν έχει αρκετά στοιχεία για να δούμε κατά πόσον το ΠΑΣ μπορεί να αποκριθεί στις ε, ανάγκες. Και όλο ένα και περισσότερα κράτη-μέλη το ζητούν. Δεν χρειάζεται συγκριματοδότηση για αυτό το λόγο και το ότι όμως είναι ανεπαρκής η διατηθέμενη χρηματοδότηση. Χρειάζονται όμως μεταρρυθμίσεις σε διάφορους στρατηγικούς τομείς. Δεν υπάρχει διαφάνεια και αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών το θεωρεί πάρα πολύ σοβαρό. Θέλουμε να υπάρξει πλήρη ενημέρωση και να δημοσιοποιηθεί η επίδοση του ΠΑΣ. Οπότε η Επιτροπή μας λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει επικύρωση του ΠΑΣ μετά το 2020 μόνο αν η αξιόλογηση καταλήξει ότι πρέπει αυτό να γίνει, ότι ο απολογισμό είναι θετικό. Και να δούμε μήπω θα υπάρξει κάποιο νέο μέσο για τι διαρροτικέ μεταφορέ. Γιατί κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε στο χάρτη πορεία στι 6 Δεκάτου του 2017. Οπότε εμεί είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί για αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις, γιατί είπαμε αυτό το μέσο φορά συνδυασμό κάποιων επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό και από ε, την ε, τεχνική αρρωγή του ΠΑΣ. Και έτσι το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κάνει μια πολιετή μεταρρύθμιση και θεωρούμε ότι η ανεπάρκεια των κονδυλίων δεν είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν ξεκινήσει οι μεταρρυθμίσεις, ότι αν ξεκινήσουν προχωράνε πάρα πολύ αργά κατά τη γνώμη μας το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις ε, υποχρεώσεων για τα κράτη-μέλη. Οπότε, ό,τι τυχόν δυσκολία υπάρξει, περιπλοκή, η η τεχνική, οι το, διοικητικές δυσκολίες, ε, όλα αυτά είναι εμπόδια αξεπέραστα. Και έτσι αυτές οι συστάσεις αναχώρα είναι θέμα το λόγιο του πολιτικού κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη με αποφασιστικότητα. Αυτά όμω η Επιτροπή δεν τα εξετάζει, έχει κεντροκατευθυνόμενη νοοτροπία. Και έτσι αφήνει έξω το παιχνίδι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ. Αυτό είναι αντίθετο στη συνδιαχείριση που επιβάλλεται από την πολιτική συνοχή από τη διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα. Αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να ισχύσει για το επόμενο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε αντιθέτω, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή για τα πλαίσια του ΣΕΦΠΕ θα πρέπει να καλύψει τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και έτσι να βοηθηθεί η εδαφική συνοχή, να υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα. Ε, γι' αυτό και η Επιτροπή Περιφερειών στην 1η Φεβρουαρίου ενέκρινε ένα ψήφισμα και απέριψε την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον κανονισμό για τα διαθωτικά ταμεία. Όσον αφορά τη χρήση του αποθέματος αυτού για να προχωρήσουμε στην άξιση του κονδύλιου προγράμματος στήριξης. Εμείς αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο είναι δόκιμη αυτή η πρόταση και αν συμβαδίζει με την ε, επικουρικότητα. Έτσι δεν θα έχουμε μεταρρύθμιση και δεν θα έχουμε και γεφύρωση των ανισοτήτων. Οπότε μας ανησυχεί το ότι εάν δεν υπάρχει συγχρηματοδοσία στην άμεση διαχείριση, α, τότε πάμε προς επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει και κάποια αντίφαση πίσω όσον αφορά την αξιοποίηση των ε, πόρων για την γενική μεταρρύθμιση και υπάρχει και συγκέντρωση θεματική όσον αφορά τα διορθωτικά ταμεία. Άρα χρειάζεται να υπάρξει τροποποίηση τώρα του κανονισμού. Αλλιώς θα έχουμε καθυστέρηση στα προγράμματα. Θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι κάποια προγράμματα θα λήξουν σε έναν μήνα από τώρα. Οπότε εμείς θα ε, μετέλθουμε την αρμοδιότητα που έχουμε σύμφωνα με το δεύτερο πρωτόκολλο για την εφαρμογή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και θα προσφύγουμε για την πρώτη της Επιτροπής ενώπιον του δικαστηρίου. Χαιρόμαστε που η αμοιβαία συνεργασία για το θέμα προχωρεί και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much for Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πολύ λεπτομερείς σας απόψεις. Ο λόγος στον κύριο Πομιέρη, συνεισηγητή για αυτό το θέμα στην ΕΟΚΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και κύριοι βουλευτές μέλη τη Επιτροπή Βουλή Ανάπτυξης. Ε, η ΟΚΕ έλαβε δύο αιτήματα διαβούλευση και εμεί επομένω ε, συντάξαμε μια γνωμοδότηση, εγώ και ο, ο, ε, ο, ο κύριος Ιβάσκο. Αυτά στις 13, 14 Μαρτίου. Και σε ανταπόκριση αυτού που ζητήσατε, με τη δική μου πνευματική λέμε ότι, θα, ότι διατυπώνονται κάποιες συστάσεις, κάποιες προτάσεις που εντάσσονται σε ένα γενικότερο όραμα και άποψη που έχουμε ως ΟΚΕ για το ότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και έτσι να έχουμε μια σύγκληση για περισσότερη σταθερότητα και ευημερία στα κράτη για τους ε, ε, Ευρωπαίους επίσης. Οπότε έχουμε το τελευταίο ανακοινωθέν τύπου της ε, ΟΚΕ, οπότε και εκεί διατυπώνουμε όλες μας τις προτάσεις για τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην είσοδο της αιθούσης μας. Όσον αφορά την πρόταση για την πρικοδότηση αυτού του προγράμματος στήριξης και σε σχέση με την προσαρμογή του γενικού στόχου, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν ε, την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης και για το ότι θα πρέπει να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών. Και όταν ληφθούν αποφάσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτό θα πρέπει να γίνει με τον κώδικα διοντολίζει την εταιρική σχέση που έχει η Ευρώπη στο πλαίσιο των ε, επενδυτικών ταμείων και ταμείων ε, διαρθρωτικών. Και έτσι να ισχύσει αυτή η αρχή, ε, οπότε και εμείς προτείνουμε κάθε κράτος μέλος να μην παίρνει πόρους εάν δεν έχει μπορέσει 100% να εμπλέξει την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την αξιολόγηση της δέσμης προτάσεων με ορίζοντα πολυετή, άρα χρειάζεται μια αυθεντική συνδιαχείριση. Ακριβώς όπως είπε και η κυρία Μάρετιτς πριν από λίγο. Το 2017 είχαμε μια πρικοδότηση 22 εκατομμυρίων και είχαμε 271 αιτήσει ε, από 17 και ζητήθηκαν 80 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ. Οπότε εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι αυξήθηκε η προοικοδότηση για το πρόγραμμα. Όμω έχουμε ακόμα κάποιε επιφυλάξει για την αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι τόσε πολλέ οι αιτήσει που έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη. Οπότε για αυτό η αύξηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει χωρίς να τεθούν να αμφιβόλο τα χρήματα άλλων ταμείων που χρειάζονται και αυτά. Οπότε συμφωνούμε με τα όσα είπε η κυρία Τόμασιτσο. Μια και επομένω η ζήτηση πιο μεγάλη από την προσφορά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορο τρόπο να μα πει τι θέλει να κάνει η αφορά την κατανομή τη νέα πρικοδότηση. Να έχει ξεκάθαρε διατάξει και στόχου για την επιλογή των μεταρρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων. Και να υπάρξουν εγγύσει για ισοτιμία μεταξύ κρατών μελών για τι πιστώσει. Και επίση θα πρέπει να μα πει ποια είναι τα κριτήρια τη επιλογή Οπότε για να χρηματοδοτηθούν οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που, που να είναι σύμφωνα με τους στόχους και τις συστάσεις για κάθε χώρα. Και θα πρέπει επίσης να υπάρξει εποπτεία όλων αυτών και αξιολόγηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο σκοπός είναι λοιπόν η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ποιότητας, να υπάρχει εγγύηση περισσότερης ανταγωνιστικότητας στον μεταπηρικό τομέα, στις υπηρεσίες και επίσης να υπάρχει καλύτερη ποιότητα στη δημόσια διοίκηση και στις κρατικές δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως, δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να στηρίζονται μόνο στην κοινοτική χρηματοδότηση όλο το θέμα της κοινωνικής ε, χρηματοδότησης στηρίζεται στην επικουρικότητα και στο ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει το καθένα να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κράτη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ. Η ΟΚΕ λέει ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις για τα κράτη αυτά, τα εκτός ευρωζώνης και θα πρέπει να δούμε αν χρειάζονται περισσότερα χρήματα επιπλέον χρήματα. Ε, πρέπει να δούμε τι ισχύει, τι προβλέπουν οι συνθήκες και τι παρεκκλήσεις ε, προβλέπονται. Θα πρέπει όμως να υπάρξει εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι άριστες ε, πρακτικές. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή ο στόχος είναι να υπάρξει μια πλατφόρμα επικοινωνίας ατουρκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Είχε σημασία για εμάς, Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως, να ακούσουμε τις απόψεις των δύο επιτροπών σας, της Επιτροπής Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ακούσαμε και τις απόψεις των συνεισηγητών. Να δούμε τώρα τι έχει να πει η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς, κυρία Μακάθη, ή κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να κάνω τα εξή σχόλια. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, την εισηγήτρια, που με την έκθεση της στηρίζει τις προτάσεις Κομισιόν. Χαιρόμαστε επίσης που μας παρέχεται μια γενική στήριξη στο έργο μας από όλους μίλησαν να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Περιορίσαμε την, τις τροποποιήσεις όσο το δυνατό περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο κανονισμός υιοθετήθηκε πέρσι το Μάιο μόλις. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος. Οπότε δεν θέλαμε να αλλάξουμε υπερβολικά το περιεχόμενό του, το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Οπότε περιοριστήκαμε μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Και ποια ήταν τα απολύτως απαραίτητα, η αύξηση του προπολογισμού στα 80 εκατομμύρια εξαιτία των αυξημένων ετοιμάτων που λαμβάνουμε και δεύτερον ένα ιδιαίτερο ποσό για τις ε, χώρες που είναι εκτός ζώνης ευρώ να τις βοηθήσουμε να ενταχθούν. Πολύ συχνά ακούμε για την ε, οικονομική ε, σταθερότητα και ισχύ, ε, ανθεκτικότητα αν θέλετε και πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες να το αποκτήσουν, να την αποκτήσουν. Ε, κάποιες χώρες κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν είχαν επαρκώς ισχυρούς θεσμούς που θα τις βοηθούσαν να ανταπεξέλθουν στην κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις ιδιαίτερα χώρες που είναι να ενταχθούν στο ευρώ να τους αποκτήσουν πριν ενταχθούν. Ευχαριστούμε για όσα είπατε για τις προτάσεις μας περί ε, στήριξη σηματοδότησης. Πολλά από όσα αναφέρατε συζητήθηκαν ήδη στην επεξεργασία του κειμένου. Η αρχή της εταιρική σχέσης της συνεργασίας, για παράδειγμα, είχε συμπεριληφθεί στην αρχή και μετά όμως δόθηκε μια συμβαστική λύση. Η δομή της προσέγγισης μας είναι προκειμένου να διαθέτουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που θα λειτουργεί σωστά. Εντός αυτού του μηχανισμού υπάρχει ένας κανόνας για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού ο κανονισμός στηρίζει τις εθνικές και τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οπότε ήδη στην αρχή πρόταση υφίστατο αυτό. Μας ικανοποιεί που μας ζητείτε να στηρίξουμε τις εθνικές κρατικές αρχές. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που και εμείς κάνουμε και προτείνουμε. Χαίρομαι που το έτοιμο αυτό υπάρχει και από τα κράτη-μέλη. Τώρα, αν χρειάζεται να δώσουμε παραδείγματα, προκειμένου να κατανοήσετε τι ενισχύσεις έχουμε δώσει με βάση τον υφιστάμενο μηχανισμό, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. Προσμένουμε σε περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμασιτς. Εισηγήτρια για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Περιμένω να συνεργαστούμε για την ολοκλήρωση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, όπως σας είπα, ε, σήμερα γίνεται η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρουσία της Επιτροπής των Περιφερειών, της ΕΟΚΕ και των σχεδόν εισηγητών. Το θέμα αυτό για μας είναι επίγον. Στηρίζουμε την κυρία Κρέιλ πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση αν θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα της. Οπότε προτείναμε το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τροπολογίες υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου, στο τέλος της μέρας, έτσι 5 το απόγευμα. Οπότε ίσως καταφέρουμε να ψηφίσουμε ψηφίσουμε στις 20 Ιουνίου. Συνεδρίασή μας στις 20 Ιουνίου. Οπότε προετοιμάστε τις τροπολογίες σας, ευχαριστούμε την συγκήτρια και όλους τους συμμετέχοντες. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που όπως σας είπα είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τις προτεραιότητες και προσεγγίσεις στη μελλοντική άσκηση της πολιτικής συνοχής. Η Παγκόσμια Τράπεζα επεξεργάζεται μια έκθεση ε, για την, ε, το ρόλο των ε, ε, περιοχών που έχουν μείνει πίσω ε, στην πολιτική συνοχή. Θα καλωσορίσω τον κύριο Μπόντεουινγκ, δεν ξέρω αν προφέρετε έτσι το όνομά σα. Όλου τέτοια λάθη κάνω με την προφορά, ζητώ συγγνώμη από τώρα. Τον Τόμας Φερόλ από την Παγκόσμια Τράπεζα. Καλωσορίσατε, αν αναγνωρίζετε τα ονόματά σα, Σας δίνω το λόγο για 20 λεπτά περίπου. Και στους δύο μαζί όμως και μετά θα διεξαχθεί συζήτηση, πιθανότατα θα σας υποβληθούν ερωτήσεις κλπ. Έχετε το λόγο. Ονομάζομαι Κρίστιαν Μπόντεβικ, μια χαρά με είπατε. Θα σας μιλήσω για την, το έργο της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από χρόνια εισαγάγαμε το, τον όρο η Ευρώπη ως μηχανή σύγκλησης. Δηλαδή εξετάσαμε όλες τις περιοχές του κόσμου και είδαμε ότι ε, η πιο γρήγορη σύγκληση στον κόσμο γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό εξαιτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, παρ' όλα αυτά έχει επικριθεί ο, όρο όρος αυτός, ή μάλλον όχι ο όρος, η ίδια μηχανή, πολλοί λένε δεν λειτουργεί σωστά αυτή η μηχανή και το ξανακοιτάμε. Η μία από ε, διαστάσεις είναι η περιφερειακή σύγκληση και συνοχή. Ο Τόμας Φερόλ συναλφόρων θα σας παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της ε, έρευνας. Η έρευνα θα δημοσιευθεί αρχές Μαΐου, οπότε μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε μερικά από τα πόρισματά της μαζί σας. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Νομίζουμε ότι προσφέρει πολλά στα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και από τη δική μας πλευρά είναι σημαντική για να, καταλαβαίνουμε, να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει με την σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο το λόγο στον συναδελφό μου τον κύριο Φερόλ. Σε ευχαριστώ, Κρίσιαν. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να αρχίσουμε με τις εικόνες. Να δούμε αν λειτουργεί. Βλέπετε εδώ βλέπετε το ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε διάφορα επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα σας ε, εκπλήξει αυτό αυτή η εικόνα βέβαια. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ανισοκατανομή που είναι φυσιολογική και σε ολόκληρο τον κόσμο και κάτι το οποίο δεν θα περιμέναμε να είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο σε όλα τα μέρη. Έχει όμως και επιπτώσεις. Επιπτώσεις στην πολιτική και κοινωνική συνοχή Έχετε δηλαδή πολύ μεγάλες διαφορές στην, στις οικονομικές επιδόσεις των διαφόρων ε, περιφερειών και για μας τους οικονομολόγους ε, φαίνεται πως έχει και συνολικές επιπτώσεις στην ε, οικονομική απόδοση. Μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των περιφερειών υπονομεύουν το δυναμικό της συνολικής οικονομικής επίδοσης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Όπως είπε ο προλαλής σας, η μηχανή σύγκληση εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσει τελευταία και δυσκολίες. Εδώ σας δείχνω σε καμπίνες την σύγκληση. Πρόκειται για συντελεστές παραλλαγών και όσο κατεβαίνει η γραμμή βλέπουμε σύγκληση. Από το 2000 μέχρι την κρίση είδαμε σημαντική σύγκληση. Η πράσινη γραμμή σας δείχνει στο επίπεδο των χωρών, πολύ σημαντική σύγκριση. Κίτρινη γραμμή, περιφερειακό επίπεδο. Όμως εκεί έληξε με την κρίση το 2008, έδειξε η σύγκριση. Τώρα αρχίζει να επανέρχεται. Δεν υπάρχουν όμω μόνο κύκλικοί παράγοντε. Η πορτοκαλία καμπύλη δείχνει μεταξύ των χωρών. Και εδώ βλέπουμε σύγκριση να συμβαίνει και μέσα στα πλαίσια της περίοδου συγκλήσεω. Μιλούμε για αστικοποίηση, τεχνολογία που συγκεντρώνει τι τις δραστηριότητες σε ορισμένες περιφέρειες και αυτό πιθανώς θα συνεχιστεί. Κάποια πράγματα τώρα ιδιαίτερα για τα οποία μιλούμε στο Growing United, στην έκθεση Growing United, θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην σύγκληση. Η τεχνολογία και εμπόριο και offshoring. Μιλούμε πολύ για την τεχνολογία, για τα ρομπότ που αφαιρούν δουλειές κλπ. Όμως αυτή η διαδικασία διαρκεί εδώ και πολύ καιρό. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες είδαμε σημαντική μείωση χειρονακτικών ε, ε, εργασιών, χειρονακτικών θέσεων εργασίας δηλαδή στην Ευρώπη και αύξηση των γνωστικών. Έχουμε και υψηλή απόδοση επιχειρήσεων που δρούν στο όριο τεχνολογίας και γνώσης. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο της τεχνολογίας και τα άτομα που έχουν τα υψηλότερα προσόντα συγκεντρώνονται επίσης σε ορισμένες περιφέρειες και αυτό θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στους στόχους της σύγκλησης. Θελήσαμε λοιπόν με την έκθεσή μας να μιλήσουμε για αυτό ειδικό στο θέμα των περιφερειών που υστερούν και μέσα στην πολιτική συνοχή τι ακριβώς γίνεται. Βλέπετε στο γράφημα δύο είδη lagging regions, περιφερειών που υστερούν. Με την πολιτική συνοχή του 2015 που και μια σχετική πρωτοβουλία με τις lagging regions χαμηλού εισοδήματο στο άνω μέρος του γραφήματος, με ιδίως στο κέντρο και στην Ανατολική Ευρώπη και άλλες που δεν προχωρούν, που δεν προοδεύουν και είναι και στο Νότο για να δείξουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά ιστορικά μεταξύ αυτών των ειδών περιφερειών και μέσα στις ε, περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος βλέπουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην οικονομική επίδοση, για παράδειγμα Πολωνία-Ρουμανία, σε σύγκριση με Βουλγαρία και Ουγγαρία. Αυτό που εκπλήσει, ε, αν δείτε τις τροχές αύξησης και τις ε, θα δείτε μια αντιστροφή μεταξύ των ε, περιφερειών χαμηλού εισοδήματο και υψηλού εισοδήματο. Δηλαδή αυτέ που είναι τώρα χαμηλού εισοδήματο μπορούν να αντιστραφούν. Και υπάρχουν δύο μηνύματα εδώ για την πολιτική συνοχή. Το ένα είναι για τι περιφέρειε εκείνε για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την παγίδα του μεσαίου εισοδήματο. Είναι σημαντικό αυτό και είναι βασικό ρόλο τη πολιτική συνοχή. Για τι περιφέρειε χαμηλού εισοδήματο σύγκριση δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο για πάντα, με τον ίδιο ρυθμό. Και η πραγματική πρόκληση για την πολιτική συνοχή στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα είναι να αποφευθεί αυτή η παγίδα του χαμηλού εισοδήματο. Να συνεχιστεί δηλαδή η αύξηση του εισοδήματο και η αύξηση τη παραγωγικότητα. Για να αυξηθεί και το εισόδημα. Κυρίω για τι περιφέρειε χαμηλού εισοδήματο. Η σημαντική πρόκληση τη παγίδα του μεσαίου εισοδήματο, Είναι να συνεχιστεί η αύξηση της παραγωγικότητα, αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ταυτόχρονα. Εδώ τονίζω κάποια πράγματα. Αριστερά βλέπετε τις περιφέρειες χαμηλή ανάπτυξη ανάπτυξης και στη μέση βλέπετε χαμηλού εισοδήματο, που ε, ε, ε, ζουν όμως μια σημαντική ανάπτυξη της παραγωγικότητας αλλά και απώλεια θέσεων απασχόλησης. όπου βλέπετε χαμηλή παραγωγικότητα, αυτή σημαίνει συμπαρασύρει και τις θέσεις απασχόλησης. Και όπως λέμε στην έκθεσή μας, είναι σημαντικό για την πολιτική συνοχή στις περιφέρειες αυτές να περάσουν οι οικονομίες αυτές σε τομείς που παράγουν για το εμπόριο και να μην ικανοποιούν μονάχα την τοπική ζήτηση που είδαμε ότι δεν αρκεί για να κρατήσει τις οικονομίες στα πόδια του στην κρίση. Πριν να προχωρήσουμε τώρα για να ξεφύγουμε από τη χαμηλή ανάπτυξη και το χαμηλό εισόδημα, πρέπει να τονιστεί ότι και τα δύο αυτά είδη περιφερειών αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ξαφνικά οι περιφερειές χαμηλού εισοδήματος πήγαν πολύ καλά η σύγκληση θα μειώσει την ταχύτητά της και αυτή είναι σημαντική πρόκληση. Έχουμε όμως και το πρόβλημα της επίδοσης των ε, αγορών εργασίας. Βλέπουμε να πέφτουν οι απασχολήσεις και στις περιφέρειες με ταχεία ανάπτυξη, χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και ιδίως γυναικών. Οι υστερούσες περιφέρειες έχουν υστέρηση κατά 10% περίπου. Αν δείτε την Ιταλία για παράδειγμα, οι υστερούσες περιφέρειες έχουν 20%, 20 μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ανοίγεται ένας τομέας εδώ δηλαδή που μπορεί να δει να ε, προχωρεί ταχύτερα η ε, παραγωγικότητα. Και το social outcome είναι πίσω από, και από την αύξηση του εισοδήματο. Και για το ΑΕΠ κατά κεφαλήν βλέπετε στον αξιοναχή. Ε, τον δίκτυ κοινωνικής πρόοδου στον άξονα ψη. Το social outcome δηλαδή υγεία, δεξιότητες, πρόσβαση σε πληροφορίες, ευκαιρίες δηλαδή για τα άτομα για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό που βλέπουμε με μοβ χρώμα εκεί τις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης όπου όχι μόνο αυτά είναι χαμηλά, αλλά ε, υστερούν κιόλα. Θα αρχίσουν να βελτιώνονται οι επιδόσεις αυτές, αλλά η βελτίωση των επιδόσεων έχει επίπτωση και στην ανάπτυξη. Και καθώς θα προχωρούμε θα δείτε ότι ο στόχος αυτός είναι σημαντικός. Όχι μόνο δηλαδή η οικονομική επίδοση ΑΕΠ κατά κεφαλή, για, να, ε, για στόχο δηλαδή για την πολιτική συνοχή. Το μήνυμα της έκθεσης για την πολιτική συνοχή ό,τι αφορά τους στόχους της είναι ότι θα πρέπει να πάνε παραπέρα από την σύγκριση του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Η πολιτική συνοχή μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική αν δεχθεί δύο στόχους. Να ενισχύσει το δυναμικό των περιφερειών και ιδίως της δημιουργίας απασχόλησης και ισότητα ευκαιριών να αντιμετωπίσει δηλαδή ένα μέτρο της κοινωνικής πρόοδου, ώστε τα άτομα όπου και αν διαβιούν, όπου και να έχουν τη βάση τους, να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες εδώ, αλλά η ιδέα του οικονομικού δυναμικού δεν είναι καινούρια. Έχει μπει στην ε, πολιτική συνοχή από την αρχή και στο προηγούμενο ε, πρόγραμμα υπήρχε και ρητά μάλιστα στο πρόγραμμα Μπάρκερ Για να γίνει το operationalizing τώρα, για να μεταφερθεί δηλαδή σε επιτόπου, εμείς έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο για να δούμε τι αναμένει κανείς να είναι η απόδοση κατά κεφαλήν αναπεριφέρεια με συγκεκριμένες ενισχύσεις ανθρώπινου δυναμικού, τοπικού και φυσικών και τομεακών. Και βλέπουμε τουλάχιστον 70% του ΑΕΠ κατά κεφαλή να προέρχεται από, αυτές τις, από αυτή τη στήριξη. Και τι αναμένουμε να δούμε σε μια περιφέρεια. Ως εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δούμε τι μπορούμε να αναμένουμε μέσα σε μια προγραμματική περίοδο, με κάποιο λόγο τρόπο. Αλλά για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να εξετάζει δύο πράγματα. Για κάθε περιφέρεια βασισμένη στην ε, πρικοδότηση αυτή να ε, ε, βοηθήσει δηλαδή στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αλλά και να στερεώσει τις, τις ενισχύσεις αυτές και για το μέλλον. Εδώ βλέπετε κάποιους χάρτες. Στον πρώτο βλέπετε το αποτέλεσμα του οικονομικού μοντέλου στο, στις πράσινες και στις πιο σκούρες περιοχές είναι με το υψηλότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ και η ΜΟΒ και οι πιο σκούρες είναι με το χαμηλότερο, όπως θα δείτε. Είναι περίπου αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Δεξιά βλέπουμε την διαφορά ανάμεσα αυτά που θα σας έλεγε το μοντέλο ότι θα έπρεπε να είναι το ΑΕΠ και αυτό που είναι. Πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο, έτσι. Αλλά είναι ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το περίπου περιφέρειες δεν εκμεταλλεύονται πλήρως το δυναμικό τους. Και αν το εκμεταλλευόντουσαν, θα αύξαναν το ΑΕΠ τους κατά 9 περίπου 100, σύμφωνα με το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πολύ ανεκμετάλλευτο δυναμικό αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, αν θέλουμε να εστιάσουμε την, τις προτεραιότητές μας για την πολιτική συνοχής, τότε οι, οι χώρες οι οποίες είναι μοβ στο δεξί πίνακα, Βουλγαρία και Ρουμανία κυρίως, είναι αυτές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Πολλές από τις ρουμανικές περιφέρειες ο, όμως επίσης θα έπρεπε να βασίσουν το μέλλον τους στην περαιτέρω εκμετάλλευση των πρικοδοτήσεων. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πίνακας για να δούμε πώς θα πρέπει να εστιάσουμε τις ενισχύσεις μας. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Αυτό που σημαίνει ως λοιπόν επανισορρόπηση των προτεραιοτήτων είναι το εξής. Το μήνυμα μας είναι η πολιτική συλλογή κάνει πολλά ιδιαίτερως εντοπισμένες, στοχευμένες επενδύσεις και σε τομιακή ανάπτυξη, ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι πέραν αυτού που θα συνεχιστεί θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε κάποια οριζόντια ζητήματα. Πέντε πιο συγκεκριμένες πολιτικές, μακροοικονομικό περιβάλλον, επιχειρηματικό περιβάλλον, ε, αστικοποίηση, προσόντα και θεσμούς και όργανα θεσμούς. νομίζω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να εστιαστεί και σε αυτά. Τόσο με χρηματοδοτικά όργανα όσο και με το συντονισμό των πολιτικών. Τελευταίες διαφάνειες ε, μιλούν για αυτές ακριβώς πολιτικές. Πρώτον, επιχειρηματικό περιβάλλον. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα σε περιοχές ε, χαμηλής ανάπτυξης ε, ε, είναι το να χαλιναγωγηθεί η μετάβαση σε μη εμπορεύσιμα. Ε, σε, σε εμπορεύσιμα, συγγνώμη. Η... Έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις που εστιάζουν σε μη εμπορεύσιμα είδη και θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιεί ε, επιχειρηματικούς δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο και είδαμε με αυτούς ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον ενδιαφέρει πάρα πολύ ακόμα και μέσα στην ίδια περιοχή, ε, σε στην ίδια χώρα, σε διαφορετικές περιφέρειες. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στα επίπεδα επενδύσεων και στα κέρδη των ε, μικρών επιχειρήσεων. Οπότε αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα. Δεύτερον, η πόλεις. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτή είναι μια, αυτός είναι ένας χάρτης της Ρουμανίας. Στο ΜΕΜΟΒ είναι η πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30.000. Ε, πληθυσμό συγκεντρώνεται στις δευτερεύουσες πόλεις και στα πρόαστια. Το μήνυμα για τις πόλεις είναι εξής δευτέρου μεγέθους πόλεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό υποεκμεταλλευόμενο ε, δυναμικό. Η πολιτική συνοχής ήδη δίνει αρκετό βάρος στις πόλεις, αλλά μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν ένα τομέα που οι πολιτικές συνοχές θα έπρεπε να εστιάσουν. Να ξεπεραστούν ορισμένες από τις τρευλώσεις που οδηγούν σε αναποτελεσματική ανάπτυξη των προαστίων, σύνδεση των πόλεων με την υπόλοιπη χώρα και μεταξύ τους, έτσι ώστε να δώσουν το δυναμικό τους. Προσόντα. Τρίτη πολιτική στην οποία επιμένουμε. Εδώ έχουμε τους δείκτες του 2012, πίσα. Ε, είναι η βαθμολογία πίσω του 2012 στις Ιταλικές ε, περιφέρειες και ορισμένες σε άλλες χώρες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και μεταξύ χωρών και μεταξύ περιφερειών. Οι καλύτερες περιφέρειες στην Ιταλία είναι στο επίπεδο των πιο προχωρημένων χωρών, ενώ οι χαμηλότερες χαμηλότερη βαθμολόγηση περιφερειών της Ιταλίας είναι στο επίπεδο των χαμηλών βαθμολογιών των χωρών της Ευρώπης. Οπότε, το μήνυμα είναι ας εστιάσουμε στα προσόντα, στην εκπαίδευση, αλλά όχι μόνο στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση. Ε, τα προσόντα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τέλος, Καμιά φορά το αποκαλούμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει αλλά σπάνια μιλάμε γι' αυτό. Τα, τα όργανα, οι θεσμοί. Οι θεσμοί συνδέονται πάρα πολύ και πολύ συχνά με την ανάπτυξη, αλλά πολύ συχνά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτούς. Το μήνυμα εδώ είναι ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεσμών και ανάπτυξη των θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, το, το, το τελευταίο που θέλω να πω σχέση με αυτό είναι ότι στην έκθεσή μας ε, ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις περιφέρειες. Όχι μόνο για τους θεσμούς, γενικά, αλλά ειδικά για τους θεσμούς. Η αλλαγή δεν θα γίνει ούτε από εμά που ε, ε, προετοιμάζουμε μελέτες, ούτε από ένα κεντρικό κράτος από την πρωτεύουσα. Η αλλαγή θα γίνει από τις ίδιες περιφέρειες, από τοπικές αρχές που θα προσαρμόσουν τις πολιτικές τους, που θα εμπλακούν άμεσα και με σίγουρα με πολύ έντονη ε, ισχυρή τεχνική συνδρομή για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ε, Νομίζω ότι η μελέτη μας ε, δείχνει ότι είναι πολλά υποσχόμενες οι ε, ε, περιφέρειες οι οποίες έχουν ένα δυναμικό να ε, αναπτύξουν. Θα είναι έτοιμη τις επόμενες, σε μερικές εβδομάδες. Growing United θα είναι ο τίτλος της. Ας αναπτυχθούμε ενωμένοι. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ναι, ίσω ναι, ίσως ισχύει αυτό που λέτε, να έχουμε ένα τέτοιο φοβερό θέμα και να μην το συζητάμε. Φάνη είναι στη λόγια και κατόπιν μάλλον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. The contribution. But when you talked about this... Uh, Ο κ. μιλάτε για τις δεξιότητες Μιλάτε για το επιχειρηματικό περιβάλλον και η δική μου εντύπωση είναι ότι οι χώρες εκπονούν κάποια προγράμματα μεταρρύθμισης για αυτό το εξάμεινο. Έχουμε την θεματική συγκέντρωση για να δούμε πώς μετρούμε τα αποτελέσματα, τη μετάβαση νέες μορφές ενέργειας κλπ. κλπ. Επομένως παραφορτώνουμε πολλά στην πολιτική συνοχή. Πέστε μας δύο λόγια παραπάνω για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. μήπως η λύση είναι να συγκεράσουμε αυτές τις προσπάθειες και να έχουμε μια τέτοια συνδυαστική προσέγγιση να είμαστε καινοτόμοι στις περιφέρειες. Δηλαδή, οικονομική πολιτική μεταρρύθμισης και περιφερειακή πολιτική συνδυασμένες. Κυρία έτσι. έχετε το λόγο. Α, μισό λεπτό συνεχίζει ο Πρόεδρος να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά σας δώσουμε το λόγο κύριε. Κυρία Μάλετη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους κυρίους από την τράπεζα. Χαίρομαι που έχουμε ακόμα μια μελέτη που δείχνει ότι η πολιτική συνοχή αποδίδει αποτελέσματα και είναι ότι είπατε ότι έχουμε κάποια γεφύρωση ανισοτήτων. Όμως, όμως, όμως, τα αναλύσατε καλά, τα παρουσιάσατε καλά ότι έχουμε μεγάλωμα του χάσματος της ε, ανισότητας μέσα στα ίδια τα κράτη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει τεχνική αρρωγή, να υπάρχει πολιτική ανάπτυξη που να σχεδιάζεται επιτοπίως και θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Μας είπε για την εξειδίκευση, την ευφυή εξειδίκευση. Είναι θέμα για κεντρικής κυβέρνησης, βιομηχανικών δυνατοτήτων, αλλά θα είναι το θέμα του πόσο συμμετέχουν οι περιφέρειες. θα πρέπει αυτή η να γίνει από τη βάση προς την κορυφή. Και να εμπλέξουμε όλους που δρούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. μικιό γεωργία, επιχειρηματίες, όλοι, όλοι όσοι ζουν σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή περιοχή, αυτοί να αποφασίσουν τι δυνατότητες έχουν και να δούμε μετά πώς μπορεί αυτά να εξελιχθούν επί τη βάση αυτής της ευφύους εξειδικευσης με κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Το πώς μπορεί αυτό συνδυαστεί με όμορες περιφέρειες κλπ. Και έτσι να πάμε για την συνοχή. Πέρα από αυτή την ερώτηση. Πέστε να κατάλαβα καλά ότι αυτό ήταν το πνεύμα των όσων μας αναπτύξε. Τώρα συμπλήρωσε στην ερώτηση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, πώς θα συνδέσουμε την περιφερειακή πολιτική με τις διαστατικές μεταρρυθμίσει, Αλλιώ δεν βγαίνει τίποτα από την πολιτική συνοχή αν δεν αλλάξει το σύστημα τη μεταρρύθμισης στο σύνολό του. Να δούμε δηλαδή πώς αυτά τώρα τα συνδυάσουμε και θα τα συνδέσουμε Ευχαριστούμε κυρία Κρέλα για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν, ε, ομολογώ ότι δεν έχω ευνηδιαστεί όταν λέτε ότι η κατάρτιση και εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας μεταξύ άλλων και για τις ιστερούσες περιφέρειες. Με ενδιαφέρει ποια είναι η θέση σας για το εξή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός ESF και EFRA για το μέλλον, για μια μελλοντική πολιτική συνοχής, ώστε να ενισχυθεί η κατάρτιση. Τι σύσταση μπορείτε να δώσετε. Και η άλλη ερώτησή μου. Είπατε ότι στις ιστερούσες περιφέρειες, lagging regions, η μη απασχόληση των γυναικών είναι σαφώς υψηλότερη από των ανδρών. Αν κατανοώ σωστά, ωστόσο, γενικά η ανεργία στις περιφέρειες αυτές είναι δραματικά υψηλότερη από τις στις άλλες περιφέρειες. χωρίς να θέλω να κάνω διάκριση ειδικά υπέρ ή κατά των ανδρών ή των γυναικών, τα γνωρίζω αυτά από την Ανατολική Γερμανία. Όταν αρχίσαμε μετά από την επανένωση των δύο Γερμανιών την προσπάθεια αναδιάρθρωσης, πολλές γυναίκες, και αυτό είναι γεγονό, πολλές γυναίκες πήγαν εθελουσίως στην ανεργία για να μην χάσουν τη δουλειά τους οι άνδρες. Γιατί οι άνδρες πιο δύσκολα δέχονται να πέσουν στην ανεργία. Δεν θέλω να γενικεύσω την παρατήρησή μου αυτή, αλλά εάν τώρα υποστηρίξετε ειδικά τις γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας, δεν θα ενισχυθεί η ανεργία. Λέτε ότι πρέπει να γίνει κάτι εκεί. Πού βλέπετε τότε ότι θα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα θα υπάρξουν μόνο αν μπορέσει να κάνει κανείς μια προσπάθεια, μια προσφορά ώστε να ενισχυθεί η αγορά εργασίας. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της ισοδύναμης ε, συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία. Προσφέρουμε να μην παρανοηθώ, αλλά θα δώσει όντως αυτό όθηση στι περιφέρειε εάν συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ κύριε Βόκοβιτς. Ορίστε έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ υψηλή η εισήγηση Είχε υψηλή ποιότητα αυτή η εισήγηση και αυτό θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας στο μέλλον. Επίσης, διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή στους επόμενους μήνες θα πρώτα να συζητήσουμε την πολιτική συνοχή, οπότε πιστεύω ότι τα όσα μας είπατε θα τα έχουμε μπροστά μας και να τα ξέρουν αυτά και αυτοί που αποφασίζουν για την πολιτική, για, τον ε, ε, προϋπολογισμό και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και για τις πλούσιες περιφέρειες και για τις λιγότερο πλούσιες. Όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη είναι πραγματικά σημαντικό κανεί κανείς να βασίζει τις προσπαθίες του επί βάση της που έχει. Να ξέρει ε, τι μπορεί να αξιοποιήσει. Γι' αυτό και είναι σημαντικό οι περιφέρειες να έχουν αρκετές αρμοδιότητες. Ε, ε, να ε, μην ξέραν ποτέ την αρχή της επικουρικότητας, αλλά πολύ σωστά θα είπατε να εστιαστούμε στις δεξιότητες, οπότε και να ενθαρρύνουμε τη, την παιδεία να βοηθήσει σε αυτές τις ε, δέουσες αλλαγές γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και ανεργίας. Διαπιστώνουμε ότι μεγαλύτερη ανεργία υπάρχει εκεί που η σχέση μεταξύ παιδείας και επιχειρήσεων είναι αδύναμη. Να μην υποτιμούμε αυτό το συσχετισμό που υπάρχει. Επίσης, όταν προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να μας δώσει ένα σωρό ε, τότε θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική συνοχή σε περιφέρειες και κράτη-μέλη. Τώρα για να δούμε κάτι άλλο να αφορά την χωροταξία και τις πόλεις. Οι πόλεις θα πρέπει να θεωρούνται ατμομηχανή ανάπτυξης. Αλλά Αλίμονα να ξεχνούμε την Ήπεθρο. Αλλήμον να ξεχνούμε το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας για την Ήπεθρο. Δηλαδή την πληροφορική, δηλαδή την ευρυζωνικότητα. Αν παρασυρθούμε και κάνουμε τέτοια λάθη, θα έχουμε χειρότερη αστιφιλία, θα μετακινούνται ακόμα περισσότεροι από τα φτωχά μέρη στα πιο πλούσια να το προσέξουμε και επίσης να κάνουμε επενδύσεις από τα Ταμεία Συνοχής εκεί όπου υπάρχει η στέρηση για την ανάπτυξη. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στις πόλεις. Τα προβλήματα θα γίνουν δυσκολότερα, θα χρειάζονται ακόμα περισσότερα λεφτά. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Να φροντίσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο επόμενος. Είναι σημαντική η γνώμη της τράπεζας για την σύγκληση. Πολλές φορές βέβαια η γνώμη της τράπεζας δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν άλλα θεσμικά όργανα. Πολλές φορές η μια τράπεζα ήταν ξεκάθαρη στο μήνυμα ότι η σύγκληση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά έχω ένα ερώτημα γιατί δεν κατάλαβα καλά τονίσατε την σημασία του ΝΑΤΣ 3 για δευτερεύουσες μεσαίες πόλεις όπως τις είπατε. Και εμείς περιμένουμε προτάσεις. ΝΑΤΣ 2 ή ΝΑΤΣ 3. Είπαμε για να 40% για τις μεσές πόλεις. Ανάλυση είναι αυτό ή πρόταση, πρόκληση να, να, να κάνουμε στροφή στην πολιτική μας. Κύριε Μπρέσο, για το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν καθιστέ να άκουσα από την αρχή τη, τη, τη, την εισήγηση. Δεν ξέρω αν το κείμενο το έχουμε έστω και ιντερνετικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να τα διαβάσουμε. Μια σκέψη και ερώτηση. Οι περιφέρειες με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης συνήθως είναι σε χώρες που έχουν ανισότητες. Στην ε, Ιταλία επίσης έχουμε περιφέρειες από τις πιο πλούσιες Ευρώπης και άλλες από τις πιο φτωχές της Ευρώπης. Οπότε όσον αφορά τις χώρες που από την άλλη μεριά έχουν ομοιογένεια και δεν έχουν μεγάλες διαφορές για την ανάπτυξη, τι γίνεται. Τι γίνεται με το εισόδημα, τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με τη γυναική πρόνοια, ε, υπάρχει ισότητα σε όλους τους τομείς, τόσο τους υποτομείς του δημοσίου τομέα και το μέσο κόστος των υπηρεσιών εφηγραμμίζονται και συντονίζονται με τις πιο πλούσιες των περιφερειών της χώρας. Εν τότε όμως η ανταγωνιστικότητα εκείνων των περιφερειών καθίσταται ε, πάντων χολή, λιγότερη. Οπότε αυτό θα πρέπει να δούμε και να δούμε και γίνεται και με τους ε, φόρους επί των ε, επιχειρήσεων γιατί υπάρχουν κάποια ε, κλασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Άρα, τι θα μας προτείνατε, γιατί αναβίβολα είναι ιστορικό το πρόβλημα. Θα το πω γι' αυτό και για την κυρία Κρέλ. Όλος ο Νότος Ιταλίας έχει πολύ χαμηλή δραστηριότητα και βασιλεύει μαύρη αγορά εργασίας. Το λένε οι στατιστικές. Όμως αυτό εν μέρη προέρχεται από διαφορετική παράδοση που έχουμε σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά αντικίνητρα λόγω της ανεργίας, λόγω της μαύρης εργασίας. Οπότε, τελικά είναι πολιτιστικό το θέμα. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένες συστάσεις ή κάποιο είδους ερεσιμότητα εξάντεκ των προτέρων. Thank Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Ο κύριος Μανσκούρ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όμως, δεν ξέρω τι γίνεται με τις προτεραιότητες για την πολιτική συνοχή. αλλά η τράπεζα έχει ως σκοπό να χορηγεί δάνεια σε χώρες που είναι στριμωγμένες και είναι υπό ανάπτυξη. Να είδα τη μελέτη σας για τη Ρουμανία, αλλά τι γίνεται με τον Νότο και για χώρες της Καρυβικής όπως η ΑΙΤ που έχουν περάσει από δυσκολίες όπως γνωρίζετε. Τι είναι πλευράς πλευρά δική σας. Και σήμερα τι θα, πού θα πάει η χώρα μετά από το σεισμό. Έχετε κάτι ιδιαίτερο να πείτε για εκείνες τις χώρες. No Βλέπω λοιπόν, να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από πλευρά των συναδέλφων. Είδατε το ευρύ φάσμα των ερωτήσεων. Α, συμπαθάτε, συμπαθάτε γιατί ο κύριος Ροπέ έχει ακόμα μια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ώρα είχα σηκώσει το χέρι μου και ζητούσα το λόγο. Τέλος πάντων, έχω κάποια σχόλια και ερωτήσεις. Η κατάσταση στα κράτη-μέλη ε, διέπεται από πολυμορφία. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο καλάθι. Αλλού υπάρχουν λίγες περιφέρειες, αλλού πολλές, αλλού υπάρχει καλύτερη ανάπτυξη, αλλού υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ιστορικές εμπειρίες. Οπότε, Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη ποικιλία όταν εμείς πρέπει να χορηγήσουμε κάποια στοιχεία. Και σας ευχαριστώ βέβαια για τα όσα μας είπατε. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα των ενεργειών σας και χαίρομαι που θεωρείτε ότι έχει φέρει θετικά αποτελέσματα η πολιτική μας συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο μεγάλη γεωγραφική περιοχή συνοχή στον κόσμο και σύγκληση σημαίνει ότι η συνοχή πάει καλά. Έχω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η δική μου χώρα, όπως και οι άλλες βαλτικές χώρες και η Μάλτα, και με ξέρετε, δεν έχουμε ε, διέρεση περιφερειακή. Αυτό για σας είναι αρνητικό ή θετικό. Έτσι φρενάρουμε τη συνοχή ή ου. Εκεί που δεν υπάρχουν περιφέρειες αναπτύσσονται οι πρωτεύουσες ταχύτερα. Και έτσι έχουμε εσωτερική ενισότητα μέσα στη χώρα δηλαδή. Πολλές φορές σε χώρες που υπάρχουν ε, περιφέρειες ε, έχουμε τριπλάσια και τετραπλάσια ανάπτυξη της πρωτεύουσα. Τι λέτε με αυτούς 800.000 Βλέπω ότι έχετε κριτήριο σύγκρισης το ΕΠ. Είναι ασφαλές κριτήριο. Για να δούμε Μία χώρα που είναι στο 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Αυτό προβλέπεται από την Ένωση. 75% σημαίνει ότι πια η χώρα, η περιφέρεια δεν είναι φτωχή. Όμως, το εισόδημα σε αυτή τη χώρα περιφέρεια μπορεί να είναι τρεις φορές κάτω από το μέσο όρο. Άρα το ΕΠ είναι ή δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κριτήριο του εισοδήματος. Γιατί για τον κόσμο μετράει το τι λεφτά έχει στο χέρι, στην τσέπη, το, το εισόδημα. Ανέφερε ήδη συνάδελφος τον ρόλο της κοινή γεωργικής πολιτικής για την σύγκληση και την συνοχή. Αυτό σας ρωτώ και εγώ για την ΚΑΠ, γιατί είναι τεράστια υπόθεση. Συνδέεται άμεσα με την υπόθεση και την γεωρευτική περιοχή που καλύπτεται από την συνοχή. Επίσης, Θεωρείτε ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να τη βελτιώσουμε, οπότε θα πρέπει να της προσδώσουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Να μην μιλάμε δηλαδή μόνο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή του θεσμικού περιβάλλοντος. Ίσως θα πρέπει να υιοθετήσουμε το πρόγραμμα Juncker για να βελτιώσουμε την συνοχή μας μια που υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη που παραέχουν πολλές ε, επιχειρήσεις. Οπότε έχουμε μόλυνση, προβλήματα για το περιβάλλον κλπ. Άρα εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έτοιμα. Για ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω υποσχεθεί, λέει ο κ. Χέτμαν, ότι θα έχω σύντομη ερώτηση. Με ενδιαφέρον άκουσα την παρουσίαση της μελέτης και την πρόταση οι περιφερειακές περιφέρειες, οι πιο απόκεντρες περιφέρειες να βελτιώσουν τους θεσμούς τους, το επιχειρηματικό τους περιβάλλον κλπ. Έχω όμως την εξή ερώτηση. Δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει, αλλά εγώ γνωρίζω πως ορισμένες περιφέρειες της περιφέρειας έχουν επωφεληθεί της ε, πολιτικής ε, συνοχής για αρκετό χρόνο και είναι ίσως το καλύτερο που τους έχει συμβεί, ό,τι καλύτερο που έχει συμβεί, αλλά αυτές οι περιφέρειες σιγά σιγά αστικοποιούνται, ενισχύουν τα προσόντα των κατοίκων τους, δημιουργούν το βέλτιστο δυνατό επιχειρηματικό περιβάλλον και στηρίζουν τους θεσμούς, τους βελτιών, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υστερούν. Έχετε καταλάβει γιατί σημαίνει αυτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, πολλές και διαφορετικές, μεγάλη ποικιλία. Έτσι κι αλλιώς θα μας ενδιαφέρει να δούμε την έκθεσή σας γραπτό, οτιδήποτε μπορείτε να μας υποβάλλετε, τις διαφάνειες να μας δώσετε, αλλά να ακούσουμε και τις απαντήσεις σα προφορικά. Ευχαριστώ. Πολύ καλέ οι ερωτήσεις. Με ξεπερνούν, δεν μπορώ σε, τόσα λίγα, σε τόσο λίγο χρόνο να τι απαντήσω. Να απαντήσω μόνο ορισμένες από αυτές. Η τελευταία ερώτηση, ότι δηλαδή υπάρχουν περιφέρειες που κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υστερούν, γιατί συμβαίνει. Ε, η διαδικασία είναι δυναμική. Οπότε, έχει σημασία το σε ποιο σημείο της πορείας σου βρίσκεσαι. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις περιοχές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, τεράστιο, με τεράστια δυνατότητα σύγκληση. Είναι εκεί ιδιαίτερα πολύ πιθανό να βλέπουμε σύγκληση περιφερειών στο μέσο όρο, αλλά ταυτόχρονη συνύπαρξη και περιοχών που υστερούν. Για παράδειγμα, οι πόλεις μπορεί να συγκλίνουν πιο γρήγορα από ότι η ύπεθρος. Μετά, Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ όλες οι περιφέρειες να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο σύγκληση. Γιατί η σύγκληση εξαρτάται και από την γεωγραφική του θέση, από την πυκνότητα του πληθυσμού τους, από πολλούς παράγοντες. Είναι μια σύνθετη συνάρτηση. Είναι μάλιστα οι δείκτες μας αναγνωρίζουν ότι κάθε περιφέρεια έχει το δικό της δυναμικό. Δεν έχουν όλες το ίδιο δυναμικό για να αναπτύξουν. Δεν ξέρω αν αρκετή αυτή η απάντησή μου. Κάποιες άλλες τώρα ερωτήσεις. Ε, κάποιες ερωτήσεις αναφέρθηκαν στις περιοχές ΝΑΤΣ 2, ΝΑΤΣ 3 κλπ. Στην έκθεση ισχυριζόμαστε ότι ένα πράγμα είναι το πώς μετριέται η σύγκληση και η ΝΑΤΣ 2 είναι ε, στάνταρ αυτό, για αυτή τη μέτρηση και άλλο πράγμα είναι η παρέμβαση που μετριέται διαφορετικά και μετριέται κυρίως σε, επίπεδο ΝΑΤΣ 3 ή ακόμα και χαμηλότερο επίπεδο. Ε, δεν μπορώ πραγματικά να συγκρίνω τις ΝΑΤΣ 2 με τις ΝΑΤΣ 3, αλλά θα πρέπει να παρεμβαίνουμε στο καταλληλότερο δυνατό επίπεδο. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι η, νάτς, η, ανάπτυξη και το υψηλό εισόδημα στις περιοχές ΝΑΤΣ 2 ε, μπορεί να κρύβουν ε, την υπόλοιπη εικόνα. Μπορεί κάτω από τις περιοχές ΝΑΤΣ 2 δηλαδή να έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε πιο τοπικό επίπεδο. Οπότε είναι σημαντικό να εξετάζουμε την πραγματικότητα σε διάφορα επίπεδα και οπωσδήποτε να ξεφύγουμε και από την ε, μέτρηση μόνο του κεφαλή Πρέπει να δούμε την ισότητα, πρέπει να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό, τις ε, δυνατότητες που δίνουν, τις ευκαιρίες, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις ικανότητες, τα προσόντα κλπ. Τώρα για το θέμα των πόλεων και της αστικοποίησης. Εδώ ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Λέμε στην έκθεση ότι οι δευτέρου μεγέθους, οι μεσαίες δηλαδή, πόλεις είναι σημαντικές, μεσαίου μεγέθους πόλεις είναι σημαντικές ε, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε το ρόλο τους όχι ανταγωνιστικά έναντι της υπαίθρου που τις περικλεί, αλλά συμπληρωματικά. Πώς δηλαδή η δική τους επιτυχία μπορεί να βοηθήσει και τις κοντινές τους περιοχές να αναπτυχθούν περισσότερο. Πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε την, τις αυτές τις πόλεις μοχλούς ανάπτυξης σε ένα πιο ευρύ γεωγραφικό περιβάλλον. Και εδώ λέμε ότι είναι σημαντική η σύνδεσή τους με υποδομές, ίντερνετ κλπ. Λέμε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και τις συνδέσεις μέσα στις πόλεις, με ηλεκτρονικές συνδέσεις κλπ, αλλά και μεταξύ των πόλεων και σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, επανέρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Λέει ότι μιλάμε για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα προσόντα, τις πόλεις κλπ. Πώς όλα αυτά συνδέονται και διαθρώνονται με την πολιτική συνοχής. Ε, όλα αυτά είναι ήδη τμήμα της πολιτικής συνοχής, η πόλη για παράδειγμα, το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε, στην πρωτοβουλία των περιοχών, περιφερειών που ιστορούν ακριβώς είχαν αναλυθεί δράσεις για να αντιμετωπιστούν κανονιστικοί, ρυθμιστικοί και άλλοι περιορισμοί που περιορίζουν ή χειροτερεύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε έχει ήδη και αυτό ληφθεί υπόψη. Το μάκρο ε, περιβάλλον, το γενικότερο περιβάλλον ε, είναι ίσως πιο δύσκολο να ενταχθεί στην πολιτική συνοχή. Για τα προσόντα... Ε, ένα από τα βασικά μηνύματα είναι ότι πρέπει να ε, συνδυάσουμε τα διάφορα εργαλεία που μας δίνει η πολιτική συνοχής. Να τα συντονίσουμε και σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα διαφορετικά εργαλεία και διευκολύνσεις που έχουμε για τον ίδιο στόχο. Αυτά. Ο λόγος στον Κρίστιαν. Thanks a lot, Tom. Ε, να εστιάσω σε δύο ζητήματα. Πρώτον, οι, γεν... πιο ευρείες μεταρρυθμίσεις ε, κοιταγμένες από κάτω στα τα πάνω. Ε, υπάρχουν κάποιοι φραγμοί ανάμεσα στο τοπικό και το εθνικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Κροατίας και της τοπικής τις ε, ε αρχές της Λαβωνίας. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η στερούσα περιοχή θα ε, αναπτυχθεί. Ιστερεί εδώ και δύο περίπου δεκαετίες. Και συζητήσεις που έχουμε με διάφορους αξιωματούχους γίνεται σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία ε, εμπόδια τα οποία έχουν σχέση με το τοπικό επίπεδο και άλλα που έχουν σχέση με το εθνικό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παράλληλα και από κοινού. Δεύτερον, για τα προσόντα. Όλοι προφανώς συμφωνούμε ότι ε, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και στα νέα προσόντα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ε, ε, επιτυχίας. Αυτό που λέμε όμως στην έκθεση είναι ότι θα πρέπει να μας αφήσει το τι για το τι περιλαμβάνεται σε αυτό όχι μόνο ενίσχυση της ε, σύνδεσης της εκπαίδευσης κατάρτισης ε, με, τον κόσμο των επιχειρήσεων και τις αγορές. Βλέπουμε πέρα από αυτό πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς αναπτύσσονται τα απαραίτητα προσόντα. Για παράδειγμα, οι νέοι που βγαίνουν από το ε, εκπαιδευτικό σύστημα και μπαίνουν στην αγορά εργασίας ε, είναι πάρα πολύ ψηλοί και έρχονται από δύσκολο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και από υστερούς περιοχές. Οπότε ένα σημαντικό βήμα είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε υστερούσες περιοχές δεν έχουν δεν υστερούν και σε βασικά προσόντα όπως ε, ανάγνωση, μαθηματικά κλπ. που θα τα βοηθήσουν αργότερα στο να βρουν δουλειά. Θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ περιφερειών και έχω την εντύπωση ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε δώσει αρκετή σημασία σε αυτές τις διαφορές. Ε, όταν εξετάζουμε τις βαθμολογίες, τις PISA, ε, συγκρίνουμε χώρες μεταξύ τους, αλλά δεν συγκρίνουν σχεδόν ποτέ τις ε, επιδόσεις ε, παιδιών που προέρχονται από ε, διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές περιφέρειες κλπ. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια ανάλυση. Τελειώνω με την ερώτηση για την ατζέντα τη σχετική με την αγορά εργασίας. Με την αύξηση της παραγωγικότητας αναμένουμε αύξηση της, απασχόλη, της δημιουργίας θέσεων και αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την εκμεταλλευτούν χωρίς φραγμούς. Πολύ συχνά υπάρχουν φραγμοί. Ακόμα και εκεί που δημιουργούνται θέσεις εργασία, υπάρχουν φραγμοί που παρεμποδίζουν κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού στο να τις αναλάβουν. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια στασιμότητα ε, όπου κανένας δεν θα βγει κερδισμένος και κανένας χαμένος. Υπάρχει περίπτωση στην ανάπτυξη κάποιοι να είναι κερδισμένοι και κάποιοι χαμένοι. Thank you. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσίαση και για την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Όλε και όλου για την συζήτηση. Εδώ ολοκληρώνει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και ίσως θα επανέλθει κάποια ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά ο εκπρόσωπο τη Παγκόσμια Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σα. Είναι πολύ σημαντικό, όπω είπα και πριν, να ακούμε από εσά να αισθανόμαστε ποια είναι η συζήτηση και τα ερωτηματικά που σα απασχολούν. Σα ευχαριστώ πολύ. το βιβλίο μας θα εκδοθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου και θα, θα φροντίσουμε να σας το ε, διαβάσουμε οπωσδήποτε και έγκαιρα. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την... Θα ζητήσω μάλλον από τη γραμματεία να είναι σε επαφή μαζί σας και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη δημοσίευσή σας. Συνεχίζουμε τώρα κυρίες και κύριοι με το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καθορισμό κοινών διατάξεων για μια σειρά από ευρωπαϊκά όργανα. Σήμερα, όπως είπα, θα γίνει η πρώτη εντολογή απόψεων. Τώρα, η αρμόδια επιτροπή είναι της περιφερειακής αναπτύξεως. Αναγκαστήκαμε να περιμένουμε λίγο για να μας πούν ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας. Έχουμε λάβει γνωμοδοτήσεις από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, μάλιστα και οι μισές, όπως ε, προϋπολογισμών, ελέγχου προϋπολογισμού, απασχολήσεως, ήτρε, τρέντ και λοιπά, καθώς και των γυναικών, δικαιωμάτων γυναικών. Όλες αυτές οι επιτροπές ενδιαφέρονται ιδιαίτερω για το συγκεκριμένο θέμα και συντάσσουν γνωμοδοτήσει. Αρχίζουμε λοιπόν με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω το λόγο στου συνεισηγητέ. ποιο θα ήθελε να αρχίσει. Εσείς κύριε Βανίστελ Ρόι. Να σας δώσω μια πρώτη εντύπωση στις και στους συναδέλφους καθώς και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το κείμενο της προτάσεως. Είχαμε και επίσκεψη του Ντομπρόσκης στην Επιτροπή μας και τον ε, παρακολουθήσαμε, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπαμε ότι υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ πολιτικής συνοχής και ταμείων συνοχής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εθνικών ε, προγραμμάτων ε, μεταρρυθμίσεων των χωρών και των συστάσεων αναχώρα. έχει ενδιαφέρον να αναζητηθούν οι μηχανισμοί που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Πρόκειται για μια δοκιμή. Το κείμενο θα γίνει ίσως και πιο εξειδικευμένο. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και με τους επόμενους κανονισμούς. Το ερώτημα είναι τι κάνουν ακριβώς. Η πλευρά της χρηματοδότησης ιδίως με απασχολεί γιατί εκεί βρίσκω ότι είναι η ίδια κατάσταση και εξακολουθώ να τελώ εν συγχύσει. Έθεσα ερωτήσει και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Του είπα, τον ρώτησα μάλλον, οι αλλαγές πολιτικής που θα εντοπιστούν στις επόμενες προτάσεις πολιτικής. Τον ρώτησα επίσης γιατί να συνδεθούν με την απόδοση. Δεν έλαβα καθαρές απαντήσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής διασύνδεση των μηχανισμών με την απόδοση. Α, μετά από τις ερωτήσεις προς τον Ντομπρόφσκης, κάναμε και μια προφορική ερώτηση ε, στην Ολομέλεια, τον Μάρτιο ήδη. Και εκεί δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο με τι απαντήσει που λάβαμε, διότι εμεί, το Κοινοβούλιο δηλαδή, με απόφαση της Ολομελία για την έκθεση Βέσφαλ, είπαμε ότι, κοίταξε πρόκειται για 21 δισεκατομμύρια και είναι αυτή τη στιγμή, ε, τα έχουν οι χώρε μέλη. Μπορεί να έχουν συμφωνήσει σε κάποιους στόχους οι χώρες μέλη. Ίσως λοιπόν να είναι σωστό να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά και πριν από το 2020. Αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Όχι, μα είπαν ευελιξία, όχι. Θέλετε να αλλάξετε κάτι στον κανονισμό, όχι, όχι αλλαγή στον κανονισμό, καμία. Τελικά είναι εντελώς ε, άκαμπτη στάση του ε, συλλογικού σώματος των επιτρόπων, της Επιτροπής στο σύνολο δηλαδή. Και έχει άλλα σχέδια. Και από την άλλη μεριά το Κοινοβούλιο έχει τις δικές του επιθυμίες. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Προτιμώ να τα πω έτσι διπλωματικά κάπως. Βέβαια δεν έχω φτάσει σε σημείο να απορρίψω όλη την ε, προσπάθεια αυτή αλλά θέλω να μάθω ακριβώ τι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο, το, το Κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο ε, να κάνει προσπάθεια και να προσκουρήσει ένα τείχο και να μένουμε χωρί απαντήσει. Να δούμε τι θα γίνει με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές προτάσεις. Ε, βρίσκομαι σε απόλυτο αδιέξοδο. Ίσως μπορεί να βοηθήσει η Κωνσταντσε Κρέλ. Ορίστε κύριε Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου φαίνεται καλύτερο να μιλήσει όχι διπλωματικά. Ας αποσύρει την πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πω διότι αυτό θα μας απαλλάξει και από πολύ περιττή εργασία. Ο κ. Βανίστερ Ρόι τα είπε πρόκειται για ερωτήσεις που έχουμε κάνει από την αρχή και δεν έχουν λάβει απαντήσεις. Και ήταν και για μένα αρκετά δυσνόητο. Ναι, σύμφωνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο. Όταν όμως έρχεται ο αντιπρόεδρος της, τον Πρόφσκης, και τα παρουσιάζει τα πράγματα αυτά, γιατί είναι αρμόδιος για την Περιφερειακή Επιτροπή και εμείς και οι δύο συνεισηγητές θέλαμε να μιλήσουμε και με τους δύο συναρμόδιους επιτρόπους και λαμβάνουμε από το προσωπικό γραφείο του Ντομπρόφσκης «Α, όχι, μια στιγμή αυτά είναι αρπρογκλησία μοντέλα της κυρίας Κρέτσου». Εγώ έχω μείνει με τα ερωτηματικά. Και πέραν αυτού, ολόκληρη η διαδικασία είναι αδιαφανής για μένα. Ο Λάμπερτ Βανίστερ Ρόι είπε ότι το performance reserve βρίσκεται ήδη στους φακέλους των χωρών μελών. Εγώ δεν γνωρίζω καμία περιφέρεια που να μην θέλει να φτάσει τους στόχους και να λάβει την performance reserve. Το γεγονός ότι δεν λειτουργεί αυτό ε, οφείλεται στο ότι έχουμε ε, εφαρμόσει με κάποια καθυστέρηση, επομένως οι χώρες μέλη δεν είναι ήδη έτοιμες. Όμως το αποθεματικό απόδοση θα πρέπει να είναι ήδη από του χρόνου έτοιμο. Αυτό θέτει όμως ένα δημοσιονομικό πρόβλημα για μένα. Έχουμε τις ετήσιες δόσεις ήδη σχεδιασμένε στην διαδικασία του προπολογισμού, στο τρέχον δηλαδή πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν προβλέπεται πριν από το 2019 να διατεθούν κονδύλια για το αποθεματικό απόδοσης. Πώς θα συντάξουν νέο κανονισμό που να πάρουν τα χρήματα, να αφαιρέσουν τα χρήματα από το Performance Reserve και αύριο μεθαύριο να χρηματοδοτήσουν πιλωτικά προγράμματα. Αυτό από όψη δημοσιονομικής πρακτικής πώς θα γίνει. Και πέραν αυτού διαρωτώ με πώς ένας νόμος ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ μπορεί να τροποποιηθεί αναδρομικά. Και η performance reserve ανεξαρτήτως του αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ή όχι, να αφαιρεθεί από τις χώρες μέλη, σε οικειοθελή βάση βέβαια σημειώνω, χωρίς να ερωτηθούν βέβαια οι περιφέρειες, παρά μόνο οι χώρες μέλη. Και εκεί η διαδικασία δεν είναι ξεκάθαρη πώς θα γίνει δηλαδή σε μια ομοσπονδιακή χώρα μέλος, πώς θα πιεστούν, πώς θα αναγκαστούν οι περιφέρειες να επιστρέψουν τα χρήματα. Όλες αυτές τις ερωτήσεις τις έθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ στην Επιτροπή μας. Μέχρι τώρα οι επιτροπές που έχω λάβει είναι, ε, οι απαντήσεις που έχω λάβει είναι μερικές ή ανεπαρκείς. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή δεν μπορούν να απαιτούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μας να πάρουμε τα 21 δισεκατομμύρια πριν από την πρόταση για το νέο ΠΔΠ και να τα επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν θα τα διαχειριστεί σε κοινή διαχείριση με τις χώρες μέλη αλλά σε central management, δηλαδή αποφασίζει μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ουσία να τους πούμε ότι α, δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά για την πολιτική συνοχή. Ενώ εμείς αγωνιζόμαστε και για το τελευταίο ευρώ υπέρ της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Δεν έχω ιδέα τι θα βάλουν στη νέα πρόταση για το ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να δώσουμε το μήνυμα και πριν από αυτό ότι είμαστε διατεθειμένε να επιστρέψουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομολογώ και το λέω καθαρά. Δεν ε, ζούμε μέσα σε μια ε, φούσκα. Από όσα ακούω δεν υπάρχει καμιά χώρα μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να λέει με ενθουσιασμό ναι εγώ θέλω, θέλω να το κάνω αυτό και ορίστε υποστήριξε κοινοβούλιο την πρόταση της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τουλάχιστον σήμερα να έχω ορισμένε απαντήσεις. Εάν δεν αποσύρει την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι να κατατηθεί η πρόταση για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δούμε, μπορεί να συμβεί αυτό. Υποστηρίζω απολύτω την πρόταση που κάνει ο Λαμπέρ Βανίστερ Ρόι να διεξαγάγουμε ακρόαση όπου να θέσουμε και το θέμα ποια είναι η στάση των περιφερειών αλλά επίσης να φέρουμε και κάποιον να μας εξηγήσει που να κατανοεί ποιε είναι οι επιπτώσει και ποια είναι η νομική κατάσταση και πώς νομικά μπορούν να το κάνουν. Και αν απαντηθούν όλα αυτά και απαντηθούν θετικά, να ερωτήσουμε τι διαδικασία μπορεί να υπάρξει. Αν είναι δυνατόν να γίνει δηλαδή τέτοιου είδου επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι τα θέματα αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί με την κατάθεση της πρότασης της Επιτροπής. Και όσο δεν απαντώνται, δεν είμαι και εγώ διατεθειμένη να επεξεργαστώ θετικές τροπολογίες και νομίζω εκεί σε αυτό δηλαδή συμφωνούμε απολύτως Λαμπέρ Βανίστερ Ρόι και εγώ. Η πρόεδρος. Ακούσαμε τους ε, συνεισηγητές και μας είπαν με λίγα λόγια ότι τα πράγματα είναι πολύ θολά. Δεν έχουν δοθεί οι απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν στην προηγούμενη συνάντηση. Αλλά ούτε προέκυψε τίποτα από την επικοινωνία μας με την Κομισιόν. Μπά και σωστό τώρα να δώσουμε τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως και απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα. Και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με τους σκιώδες συζητητές. Γιατί Προς το παρόν υπάρχει αυτή η πρόταση για την ε, ε, έκτακτη ακρόαση των δύο συνεισηγητών και μετά την ε, παρουσίαση νομίζω ότι οι πάντες θα συμφωνούν ότι χρειάζεται αυτή η εκτακτή ακρόαση. Για να δούμε τώρα τι απαντήσεις μπορεί να προγύψουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώ με τον κύριο Φων Μπρέσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές που υπέβαλαν παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Δεν μπορώ να σας απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, αλλά να προσπαθήσω λίγο να σας διαφωτίσω για την πρότασή μας. Νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να τονίσει το πόσο σημαντικέ είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί το ξέρουμε όλοι, αλλά τελικά Αυτά τα μέσα πολιτικής διατυπώνονται στην πρότασή μας θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποια ευκαιρία. Και έτσι τα κρατημέλη σε βάση εκούσια και θελαντική μπορούν να προχωρήσουν εάν θεωρούν ότι είναι σωστό. Χρησιμοποιώντας αυτό το αποθεματικό επίδοσης και απόδοσης όλο οι εν για να κάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε αυτή την επιλογή στα κράτη-μέλη. Γιατί ίσως έχουμε κάποιες καταστάσεις κατά τις οποίες τα προγράμματα δεν θα πετύχουν τα δέοντα και για να μην χάσουν τους πόρους τα κράτη-μέλη μπορούν να τους αξιοποιήσουν μια που δεν τους τα πάρει κανείς αυτά τα χρήματα δεν θα τα ανακτήσει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσουν επομένως αυτά τα χρήματα για άλλους σκοπούς και στόχους άρα να προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία στα κράτη-μέλη δεν θα αναγκάσουμε κανένα κράτος καμία περιφέρεια έτσι λειτουργεί το σύστημα Οπότε αυτά θα βγουν από τα προγράμματα. Θα έχουμε αυτή τη δέσμευση για τη μεταρρύθμιση, αλλά η εταιρική σχέση των περιφερειακών εταίρων ε, θα περνάει μέσα από μια διαβούλευση, μέσα από μια συμφωνία για αυτή την μεταβολή. Αλλιώ δεν γίνεται τίποτα γιατί βέβαια οι διατάξει, βασική αρχή της και πολιτικής συνοχής είναι ότι αυτά αυτές οι αρχές, αυτή η εταιρική σχέση, ε, αυτή η συνεργασία για το πρόγραμμα θα πρέπει να ισχύει. Επίσης, όλα αυτά θα μας διαφωτίσουν για την περίοδο 2020, μια που και εκείνη την περίοδο θα δρομολογήσουμε ένα εργαλείο παρόμοιο. Άρα, μπορούμε να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα με τις επαφές, τις διπλωματές, με μίλη για τα είδη των μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαμε να στηρίξουμε. Πώς θα θέσουμε κάποιους σκοπούς και στόχους. Οπότε, γι' αυτό σας λέω ότι θα βοηθούσε. Εάν πριν το 2021 αρχίσουν να ισχύουν το, τα πολιτική δημιουργικά πλαίσια ή το πλαίσιο τέλο πάντων, να έχουμε πιλωτικά διαφωτιστεί με αυτό το εργαλείο που συζητούμε. Άμεση διαχείριση, είπαμε. Και πιστεύουμε ότι στη σημερινή συγκυρία είναι μικρότερο το ρίσκο. Εάν έχουμε τους κανόνες για τη συνδιαχείριση. να σκεφτείτε ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος θα είναι, ε, ποιος έχει την, την, ε, κυρίως για τη διαχείριση, όλα, όλα αυτά πρέπει κανένας να λάβει υπόψη. Αν δεν να κινηθεί στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, ούτε τίποτα μας απαγορεύει στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, να εφαρμόσουμε εν μέρη την ε, συνδιαχείριση. να σκεφτείτε την πρωτοβουλία για τις πόλεις που διαχειριζόμαστε έμεσα. Άρα τα κονδύλια συνοχής, αυτά τα χρήματα δεν είναι υποχρεωτικό να περάσουν από συνδιαχείριση. Αυτή την προσέγγιση διαλέξαμε. είναι τα πράγματα απλά. Και γι' αυτό και πρώτη προτείναμε τέτοιου τους διαχείριση. Ούτε θα πάρουμε πόρους που είχαν διατεθεί το 2019, θα διαθέσουμε αλλού. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας επισημάνουν κατά το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, για τις μεταρρυθμίσεις του 19 ότι θα υποβάλουν τον επόμενο χρόνο τα κράτη-μέλη. Θα είναι μια ευκαιρία να επισημανθεί από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή το αν θέλουν να μετέλθουν, να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία. Και μετά θα δούμε μας ποιοι είναι οι στόχοι, τι δεσμεύσεις θα υπάρξουν και επίσης θα δούμε τι θα αποφασίσει το κράτος μέλος, γιατί αυτό θα αποφασίσει. Τι θα εισφέρει ως προσπάθεια, ως πόρος για τη δέσμευση που θα αναλάβει. Όλα αυτά θα γίνουν όσο επιτοπλίσουν το πρώτο Ξένο του 19. Πυρωτική προσπάθεια. Είναι αυτή θέλουμε να είναι σύντομη, θέλουμε να είναι απλή. Και γι' αυτό και η περίοδος εφαρμογή θα καλύψει μόνο τρία χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι οι ρυθμίσεις συνήθω παίρνουν περισσότερο χρόνο. Είναι το θέμα βέβαια της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, αλλά δεν θα περάσουν από αξιολογήσεις. Γιατί αυτό δεν θα είναι πιλωτική προσπάθεια που, όπως είπα, θέλω να είναι απλή και πιλωτική. Να είναι μια επιλογή για να τα κράτη-μέλη. Τελευταίο αλλά σημαντικό, έχω να σας πω ότι ήδη έχουμε την Πορτογαλία. Ήδη επεσήμενε στην Κομισιόν ότι θα ενδιαφερόταν να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Άπαξ βέβαια και οι συνομοθέτες συμφωνήσουν για τις προτάσεις της Κομισιόν και θεσπίσουν ε, το σχετικό νομοθέτημα εδώ βάζουμε τελεία και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Και τώρα, θέλει τον λόγο ο κύριος ή κυρία Τζενόριο από την Κομισιόν. Όχι. Δεν θέλετε, δεν θέλετε. Καλώς, λέει η Πρόεδρος. Και συνεχίζουμε τώρα την ε, τακτική διαδικασία με τους σκιώδεις εισηγητάς. Τόμασιτς. Η ομάδα του ECR δεν αμφισβητεί την ανάγκη να στηριχθούν οι διασωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αμφιβάλλουμε σοβαρά για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν. Για να εισαχθούν ε, η εισαγωγή αυτών των αλλαγών τώρα με τις παρούσες δημοσιονομικές πρακτικές ε, θα απορριθμίσει πάρα πολύ την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ε, πολιτικής συνοχής και ταυτόχρονα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής γιατί θα πρέπει να μετακινηθούν κονδύλια για να υποστηριχθούν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ε, διενεργούνται εκτός της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει η Κομισιόν να ε, χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα αποθεματικά ε, επίδοση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα δημιουργηθεί ο κίνδυνος, μάλιστα, ο μηχανισμός να μην προλάβει να ε, δοκιμαστεί επαρκώς στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, κάτι που θα οδηγήσει σε προβλήματα και στο μέλλον. Η, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνει με, τα... με τους στόχους που είχε. Ευχαριστώ πολύ, ο Βαν Μίλτεμπερκ. Νομίζω ότι οι διαφορετικές αλλαγές ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές αλλά θα πρέπει να θέσουμε σοβαρούς όρους για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Η θέση της ομάδας μας θα εξαρτηθεί από τις διευκρινήσεις που θα μας δώσει η Κομισιόν στα ερωτήματά μας. Κοίταξα την πρόταση. Βλέπω στο καινούριο άρθρο 23 ότι η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια πρόταση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη και τα ποσά που θα δεσμευθούν από τα αποθέματα επιδόσεων για αυτούς τους στόχους με βάση ποια κριτήρια. Δεν θα αντιμετωπίσουμε σε ένα-δύο χρόνια προβλήματα με το ελεγκτικό συνέδριο αν δεν εφαρμοστούν κριτήρια, αν δεν χρησιμοποιηθούν κριτήρια. Πώς θα ε, υπολογιστούν τα ποσά. Τα ποσά δεν συνέονται με το κόστος. Δεν συνέονται με τα κόστη. Ή μίλησατε για την Πορτογαλία. Τι ακριβώς θέλετε να χρηματοδοτήσετε. Δεν θα πρέπει να έχετε κριτήρια τα οποία να είναι γνωστά. Δεν θα ξέρουν όλοι ποια είναι τα παραδοτέα, σε ποιες χρονικές στιγμές. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για μικρής διάρκειας ε, Παρεμβάσει. Πρέπει να πάρουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν είναι να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Αν αυτό πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα ε, και αποτύχει, τότε μετά πώς θα το επαναφέρουμε μετά το 2020, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το αποθεματικό επίδοσης υποτίθεται ότι θα ήταν κίνητρο. Τώρα τι, θα χαλαρώσουν όλα τα κράτη-μέλη και θα πούνε ότι αφού δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις προτεραιότητές μας, α, θα το χρησιμοποιήσουμε σε ένα χρόνο, λίγο αργότερα, τουλάχιστον εν μέρη για άλλα πράγματα. Δεν θα επικρατήσει χαλάρωση. Το αποθεματικό αυτό, απόδοση, επίδοση, θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο. Και έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη στιγμή. Ε, είναι επίγον όμως να απαντηθούν. Η θέση μας εξαρτάται πάρα πολύ από τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η πράσινη. Όχι. Κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτέλους μετά από πέντε μήνες φτάσαμε στο σημείο να συζητούμε την πρόταση της ε, Κομισιόν. Θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για απλή τροποποίηση του κανονισμού των κενών διατάξεων. Είναι απόδειξη του τι ρότα θέλει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή για τη συνοχή. Οπότε μακάρι να είναι ενωμένα και αποφασιστικά τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Οπότε αυτό το αποθεματικό τώρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε τώρα έχουμε συνδυασμό των πέντε διορθωτικών ταμείων. Η Ιταλία μετά την Πολωνία έρχεται δεύτερο όσον αφορά την ωφέλεια από τη συνοχή. Μιλούμε για 2,5 δις από το συνδυασμό της βοήθειας. Ε, των 5 ταμείων 14 με 20. Υπάρχουν διάφορες καινοτομίες σε σχέση με τους παλιότερους κανονισμούς. Είναι πιλωτική φάση, όπως είπε η Κομισιόν, για να έχουμε ένα delivery tool, να έχουμε ένα εργαλείο και να φτάσουμε στη μεταρρύθμιση και από την επόμενη χρήση ε, ή την περίοδο 21-27 να μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη πρικοδότηση Είπατε ότι θα πρόκειται για κάτι το εκούσιο ε, σε σχέση με το αν θέλουν τα κρατημένα να πάρουν τους πόρους, αλλά θα πρέπει όλα αυτά ε, να τα συμφωνήσουν σε εισαγωγικά τα κρατημένη με την Κομισιόν να υπάρξει συντονισμός των οικονομικών πολιτικών να λάβουν υπόψη επίσης το σκοπό τα όσα αποφασίστηκαν για την Ευρωζώνη το Δεκέμβριο του 2017 και με τους κοινωτικούς κανόνες να αναβαθμίσουμε τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, να αναγκάσουμε τα κρατημέλη να κάνουν τις αναγκαίες θεωρηθήσεις μεταρρυθμίσεις, απασχόληση, παιδεία και δικαιοσύνη επίσης. Τα έχουμε πει επανειλημμένα. Βεβαίως και συμφωνούμε για τις μεταρρυθμίσεις και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και ό,τι άλλο υπονομεύει το κράτος προνοίας. Γιατί όμως να παίρνουμε πόρους από την συνοχή. Συμφωνούμε. Γιατί αυτό είναι ένα από τα πολλά χτυπήματα που έχουν δοθεί στην συνοχή. Καλά, έχουμε τη συνοχή για τα κατεπήγοντα, όμως αυτό τώρα πάει κόντρα σε ό,τι προβλέπουν οι συνθήκες, στο πνεύμα των συνθήκων για την συνοχή. Οπότε έτσι ανατέλει ένας, φαίνεται ένας κίνδυνος. Τι θα γίνει με αυτούς που δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα ταμεία επί τη βάση των επιδόσεών τους. Υπάρχουν χρήματα στα αποθεματικά. Εμείς θα κατεβάσουμε τροπολογίες μόλις οι συνεισηγητές μας παρουσιάζουν το σχέδιο κειμένο τους. Ε, ευχαριστούμε λέει πρόεδρος. Ακούσαμε τους συνειδητές των πολιτικών ομάδων, τώρα έχουμε άλλα δύο μέλη από τους συναδέλφους της ε, Ρέτζη που θέλουν να λάβουν το λόγο και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, ΟΚΕ για να μας παρουσιάσει την άποψή της όσον αυτό το θέμα. Κύριε Νόβακο, έχει το λόγο. Thank you very much. I'm not expert on communication. Ευχαριστώ. Δεν είμαι ειδικό στην επικοινωνία ούτε στις δημόσιες σχέσεις, αλλά θέλουν, θέλουν περισσότερα στοιχήματα οι συντονιστές, να θέλουν βοήθεια για να αποφασίσουν ίσως κάτι από την επικοινωνία μας βοηθήσει. Ήδη από τότε που ξεκίνησε τη διαδρομή της ε, αυτή η νομοθεσία είπαμε ξεκινήσαμε με 140 εκατομμύρια για το SRSP. Και πολλοί συνάδελφοι ήταν επιφυλακτικοί για το πώς τα 5 εκατομμύρια μέσο όρο μέρο θα μπορούσαν να αποδώσουν για τι δραστηριοτικές μεταρρυθμίσεις. Μετά, η αυξήθηκε και τώρα έχουμε την παρούσα πρόταση έστω για αυτή την περίοδο που προβλέπεται σύντομη. Δεν μπορώ να κάνω τώρα αξιολόγηση και περιμένω πρώτα-πρώτα να κρίνουν το θέμα οι συνεισηγητέ, αλλά ευθύ εξ αρχή Θα πρέπει να σκεφτούμε τελικά αν θα γίνει βήμα πρόοδου. Τους τρεις τελευταίους μήνες ο κόσμος με ρωτάει ασταμάτητα και τι θα γίνει με τις επιδόσεις, την απόδοση, τι θα θέλετε να παραλύσει. Τι να τους πω. Και για τις κοινέ διατάξεις τελικά όσον αφορά τους δικαιούχους δημιουργήσαμε περιβάλλον ανασφάλειας. Είχαμε το CPR, μετά είχαμε το αποθεματικό των επιδόσεων, μετά είχαμε το performance delivery. Αλλάζουμε κάθε τόσο το, το, το, την νομοθεσία που διέπει τα ταμεία. Ε, απλουστεύσουμε τις ε, κινήσεις μας. Έτσι θα χτίσουμε εμπιστοσύνη και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον και του συμφέρον των α, δικαιούχων. Αλλιώς θα πρέπει ασταμάτητα να κάθομαι και να εξηγώ στις ΜΜΕ, στους, στους Δήμους και στις κοινότητες ε, γιατί αλλάζουμε κάθε τρεις και λίγο την νομοθεσία. Μάλιστα, ναι, είναι πολύ σημαντικό να απαντηθεί το ερώτημα του τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Εντάξει αφού έχουμε αυτό το αποθεματικό επιδόσιο για να συμπληρώσουμε την τεχνική αρρωγή της συνοχής και αν αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις ενισχύσουμε την εξειδίκευση, την και κλπ. Και με μια τέτοια μέλουσα πολιτική συνοχή, εντάξει, θα δώσουμε το πράσινο φως. Και φυσικά συμφωνούμε μια που είναι εκούσια μέτρα αυτά. Είπατε όμως ότι θέλετε αυτό να το διασυνδέσετε με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Εμ τότε αναδύονται κάποιες αμφιβολίες, γιατί άμα κάνετε αυτή την διασύνδεση, τότε πάμε σαν ένα νέο SRSP. Μα τα είπαμε, τα είπαμε στην αρχή της συνάντησης. Σήμερα. Μα τι φτιάχνετε ένα SRSP μέσα στην πολιτική συνοχής και ρίχνεται μέσα και το, το αποθεματικό επιδόσεων. Μα τα είπαμε. Δεν είναι σωστό να περάσει από συνδιαχείριση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για την ε, υλοποίηση. Με άμεση, κατευθείαν διαχείριση θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι κι άλλο πει. Αυτό να έχουμε κατά νου. Και επίσης είπατε τώρα θα πριτανεύσει η ευελιξία ωραία όποτε ο καθένας μπορεί να επιλέξει πώς θα ξοδέψει τα χρήματα στις μεταρρυθμίσεις. Όμως έχω τα κρατημέλη, χτυπάνε πόρτα της Κομισιόν και λένε επιλέγουμε πόρους, ας πούμε για πολιτιστική κληρονομιά, για αναπτυξιακά σχέδια. Και έχω συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί στην Κροατία απροβήσαμε 100% για αυτή την προτεραιότητα του πόρους. Όμως τώρα δεν θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε, να κάνουμε μεταφορά των πόρων για άλλη προτεραιότητα. Ναι, τα χρειαζόμαστε τα χρήματα, αλλά πού είναι η ευελιξία, δεν υπάρχει τώρα. Πού είναι η ευελιξία αν εξαναγκάζονται τα κράτη-μέλη για τους σκοπούς που επιλέγει η Επιτροπή. Άρα, γι' αυτό προβληματιζόμαστε. Πού το πάτε, τι θέλετε να πετύχετε σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλοι συνάδελφοι της Ρέτζη να θέλει το λόγο. Όμως θα δώσουμε την σχετάλια στον κύριο Παλνιέρη για να μας πει τα της ΟΚΕ για το θέμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για την ΟΚΕ είναι μεγάλης ε, σημασίας το να έχουμε ένα τέτοιο μέσο για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε να τηρηθούν τα όσα έχουν υποσχεθεί τα κρατημέλη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για άλλη μια φορά όμως, τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να εξευρεθεί ένας ορισμός τι εστί διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Οπότε γι' αυτό και σας επισημαίνουμε ποιες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν σε αυτή την σύντομη περίοδο να οδηγήσουν σε περισσότερες δημόσιες δαπάνες και θα μπορούσαν επίσης πιο μακρόπνο να αποδώσουν περισσότερο. Τα θεσμικά όργανα επομένως θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τα κρατημέλη ούτως ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερη ολοκλήρωση, περισσότερη σύγκληση στην Ένωση. Ε, γι' αυτό και εμείς δίνουμε το πράσινο φω. Να υπάρξει αυτό ο μηχανισμός, να είναι κίνητρο για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και να έχει το, τη δική του αυτόνομη χρηματοδότηση στα πλαίσια του πολιτού δημοσιακού πλαισίου. Εμείς βέβαια θεωρούμε ότι αυτά ισχύουν ε, γιατί είναι προσωρινή αυτή η λύση της Κομισιόν. Είναι πιλωτική προσπάθεια και στηρίζεται σε αυτό το αποθεματικό επιδόσεων. Αλλά βέβαια ε, πάλι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση εάν οι παρεμβάσεις γεφυρώσουν την οικονομική ανισότητα και αυτό κοινωνικά βιώσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει επιμελής δυναμική εποπτεία για το τι γίνεται κατά αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Για αυτό και εμείς επαναλαμβάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει, να ισχύει και να εφαρμοστεί η αρχή της εταιρικής σχέσης, της εμπλοκής επίσης των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και αυτοί να εμπλακούν σε όλη την διαδρομή και στην υποπτία και στη διαχείριση και στην στρατηγική αξιολόγηση αλλά και στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων, επεμβάσεων τέλο Ευχαριστούμε πρόεδρε, ευχαριστούμε τους συνεισηγητές που είναι πρόθυμοι να έχουμε διμερείς επαφέ. Τώρα έχουμε την πρώτη από τις πολλές προσφέρουμε σε ευκαιρίες τόσο ώστε να έχουμε σε τακτά διαστήματα συνεργασία για τα θέματα αυτά της κοινού ενδιαφέροντος ημών και ημών. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να απαντήσετε ως μέσα από τις ερωτήσεις ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω σε τρία ζητήματα. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε πιο σαφείς, γιατί δεν λέμε εξ αρχής ποια είναι τα κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα αξιολογήσουμε τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Γιατί ενδεχομένως έχετε την εντύπωση ότι εμείς ιδιοποιούμε θα κάποια εξουσία. Ο λόγος για τον οποίο δεν το κάνουμε είναι γιατί δεν γνωρίζουμε τι είδους μέτρα και τι είδους μεταρρυθμίσεις θα εγκρίνουν ή θα προτείνουν τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, αναφέρθηκα στην Πορτογαλία προηγουμένως. Οι πορτογαλικές αρχές θέλουν, για παράδειγμα, να εξετάσουν πώς μπορούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα διαβίου κατάρτισης. να, με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, μια συγκεκριμένη πρόταση. Θα μπορούσαν όμως να ε, προτείνουν προ... μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, του ε, επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλπ. Είναι πολύ δύσκολο εκ των προτέρων λοιπόν να δηλώσουμε εκ των προτέρων πώς θα αξιολογήσουμε τα μέτρα που θα προταθούν. οι προτάσει είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν δεν πρόκειται να πει να το ποσό, να, πια, είναι το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που περιμένουμε από τα κράτη-μέλη είναι αυτά να μας υποβάλουν μια πρόταση, να μας πούνε τι θέλουν να, ποια μέτρα θέλουν να εφαρμόσουν, ε, να μας ζητήσουν τα κίνητρα, να μας καθορίσουν τους στόχους, τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα. Και εκεί θα διαπραγματευτούμε. Δεν θα το επιβάλλουμε εμείς όμως. Και μετά, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς την έγκριση των ίδιων του των περιφερειών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, που την ξέρω καλύτερα. Αν θέλει, να, αν θέλει μια η χώρα να μετακινήσει κάποια ποσά από το απόθεμα για τη Βαβαρία, για την κάτω Σαξονία κλπ. Οι περιφέρειες θα πρέπει να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να το, το κράτος να πάρει τα λεφτά και να τα διοχετεύσει αλλού. Δεύτερον, γιατί δεν χρησιμοποίησαμε την, τα όργανα πολιτικής συνοχής για να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Για τον λόγο του ότι η πολιτική συνοχής εστιάζεται μόνο στι επενδύσει. Μερικέ μεταρρυθμίσει πράγματι χρειάζονται, ε, χρειάζονται επενδύσει. Για παράδειγμα, μεταρρύθμιση στην αγορά εργασία που χρειάζεται ε, ε, επανεκπαίδευση ε, κλπ. Αυτό, ναι, αυτά είναι μέτρα που χρειάζονται επενδύσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα που είναι πιο διοικητική ή ρυθμιστική φύση. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να υπολογίσουμε το κόστος μιας επένδυσης, μιας μεταρρύθμισης, συγγνώμη. Οπότε η προσέγγιση μας είναι να πούμε θα χρησιμοποιήσουμε μια καινούρια δυνατότητα του κανονισμού Omnibus και η πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά τι έγινε τότε που είναι οι πληρωμές έναντι όρων Οπότε εκεί δεν επιστρέφουμε ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί μέσω τιμολογίων κλπ. Τίθενται στόχοι, μπαίνουν όροι και η εκπλήρωση αυτών των όρων οδηγεί στην πληρωμή. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης από ότι η πολιτική συνοχής που βασίζεται στην ε, επιστροφή συγκεκριμένου κόστους, είτε είναι υπολογισμένο είτε είναι πραγματικό. Τέλος, γιατί θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να το συνδέσουμε με τα εθνικά προγράμματα ε, ε μεταρρυθμίσεων. Γιατί το ευρωπαϊκό εξάμεινο έχει σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και είναι λογικό να χρησιμοποιούμε ένα υπάρχον πλαίσιο όχι μόνο για να προτείνει το κράτος μέλος μεταρρυθμίσεις, αλλά και προκειμένου η Κομισιόν να παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν εκδίδει ανά χώρα εκθέσεις και συστάσεις. Εκεί θα υπάρχει μια, ένα κεφάλαιο που θα αναφέρουμε αν βλέπουμε πρόοδο στις δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα ήταν φυσιολογικό να δημιουργήσουμε ένα καινούριο διαφορετικό σύστημα αφού έτσι κι αλλιώς υφίστανται αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά. Αυτή είναι η λόγη. Thank you very much, Mrs. Krell. Mr. Ευχαριστώ, κυρία Κρέλ, Μάλιστα, κυρία Κρέλ. Δεν με πείθουν πολύ όλα αυτά και ούτε θα εκπλαγείτε που το λέω. Κύριε Φον ε, θυμάστε ότι ούτως ή άλλως το Κοινοβούλιο δεν ήθελε αυτό το αποθεματικό επίδοση, το οποίο δεν είναι πραγματικό αποθεματικό επίδοση, διότι η στόχη είναι τόσο χαμηλή που ήδη προ όλοι εδώ συμφωνούσαμε ότι κάθε χώρα μέλο θα καταφέρει να επιτύχει του στόχου. Το ξέρετε αυτό άλλωστε. Εσείς διατυπώσατε τους στόχου αυτούς σε συνεργασία μαζί μα. Δεν μπορώ λοιπόν να αντιληφθώ γιατί σε τούτο εδώ το χρονικό σημείο αποφασίζουμε χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική συνοχή τα δαπανούμε για άλλα πράγματα. Ασφαλώς σημαντικά πράγματα. Και εγώ θέλω να γίνουν διαφθορτικές ε, μεταρρυθμίσεις όμως αυτό δεν είναι ο στόχος της πολιτικής συνοχής. Εγώ εδώ οφείλω να υπερασπιστώ την πολιτική συνοχής. Να υπερασπιστώ τις περιφέρειες εκείνες που έχουν ιδέες και project για να ε, φέρουν, να εξισώσουν, να ε, απομειώσουν τις διαφορές μεταξύ, τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Αυτά τα λέει και η συνθήκη. Έρχεται όμω τώρα η Επιτροπή και λέει «Α, θα σα πάρουμε πίσω 21 δισεκατομμύρια». Βέβαια, σε οικειοθελή βάση. Στη Γερμανία δεν πρόκειται να βρείτε πλειοψηφία μεταξύ των ομόσπονδων ε, κρατηδίων. Εγώ ρώτησα από εδώ και από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν. Η Γερμανία χρησιμοποιεί άλλωστε τον μηχανισμό SRSP. Υπάρχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων και στη Γερμανία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εκεί δεν γίνεται τίποτα από μεταρρυθμίσει. Τώρα, Εάν είχατε καταθέσει πρόταση τι ενδεχομένως μπορεί να γίνει με μη απορροφηθέντα ε, κονδύλια της performance reserve ή με άλλα κονδύλια από εδώ και από εκεί, τι θα μπορούσε να γίνει εάν για παράδειγμα ε, δαπανόταν για στόχους συνοχής σε άλλες περιφέρειες ή εάν υπεστήριζε κανείς έξτρα κάποιες ε, περιφέρειε που θα είχαν πάει καλά, κάτι που θα ήταν πραγματικό αποθεματικό επίδοση. Δεν θα ήμασταν εδώ τώρα να μαλώνουμε, αλλά να τα βγάλετε όλα αυτά εκτό και να προσπαθήσετε να οργανώσετε κάτι το απολύτω διαφορετικό, θεωρώ πάλι εδώ ότι δεν, δεν ε, έχουν απαντηθεί επαρκώ οι ερωτήσει μου. Επιμένω, θα ήθελα να γίνει ακρόαση. Και δεύτερο, δεν αντιλαμβάνομαι, δεν θεωρώ δηλαδή ότι το βήμα αυτό είναι σωστό, τουλάχιστον επί της παρούσης. Ευχαριστώ κύριε Πανίστρε Ευχαριστώ. Δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα να πω. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα από την πρόταση εννοώ, λέει ο κύριος Βανίστερ ε, Υπάρχει ένα θέμα. Το Κοινοβούλιο θέλει να τροποποιήσει την CPR και αν όχι, το ανάποδο από αυτό που λέει η κυρία Κρέλ. Δηλαδή η Κομισιόν μπορεί να τα αποσύρει τα χρήματα, χωρίς να σημαίνει ότι χάνονται αυτά, διότι ενσωματώνονται στις προτάσεις του Ιουνίου. Τίποτα δεν χάνεται. Πρόκειται για γνώση, η οποία δεν ε, υφίσταται κυρώσεις. Αν δεν υπάρχει γνώση αυτή, τότε να πάμε για γνώση. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να πω ότι το επόμενο βήμα μας θα είναι η συζήτηση για το σχέδιο εκθέσεως για το νομοθέτημα. Όμως σήμερα οι δύο συνεισηγητές, επίσης και όδης, ζητούν περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη επιβεβαίωση και επισημαίνουν ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Βον Ήταν ε, πολύ καλή η προσπάθειά του, αλλά προφανώς δεν ικανοποίησατε το κοινό σας. Δεν θα κλείσω λοιπόν τη συζήτηση εδώ με υπόσχεση για σχέδιο εκθέσεως, αλλά σήμερα στην διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών θα συζητήσουμε το ενδεχόμενο διενέργειας ειδικής ακρόασης, διότι όταν υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις χρειαζόμαστε περισσότερες απαντήσεις. Ας κλείσουμε τη συζήτηση λοιπόν εδώ για το θέμα αυτό για σήμερα και θα συνεχίσουμε αργότερα με τους συντονιστές. Αυτό και το τελευταίο θέμα τη σημερινή διάταξη για σήμερα. Να συνεχίσουμε αμέσω με τους συντονιστέ. Ωραία. Λοιπόν, τότε, τα πρόσωπα που δεν συμμετέχουν ε, στη συνάντηση των συντονιστών, ας αποχωρήσουν. Ευχαριστώ.